Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας καλωσορίσω σε αυτή την ειδική αίθουσα. Δεν ξέρω γιατί είμαστε εδώ. Εδώ είμαστε πάντως. Δεν σας βλέπω καν. Χρειάζομαι γυαλιά για να μην πω τηλεσκόπιο να σας βλέπω. Τέλος πάντων, σας καλωσορίζω. Έχετε ερωτήσεις για την ημερησία διάταξη, όχι. Ούτε ανακοινώσει έχω εγώ. Πάμε λοιπόν μέσα στο σημείο 3. Προτεραιότητα στον τομέα των υγειακών υποδομών. Ο συνάδελφος ο Ζαβάκνερ είναι ο εισηγητής μας. Τον είδα, πού είναι, α, να, εκεί, εκεί είναι ο υπεύθυνο εισηγητής και δεν θέλω να του δώσω το λόγο αμέσω. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ας προσεγγίσουμε την ανάλυση του εγγράφου εργασίας που έχω την τιμή να παρουσιάσω ενώπιον αυτών συναδέλφων ευρωβουλευτών. Καταρχήν να επιμείνω για το ότι οι στόχοι μας για την ενεργειακή πολιτική των ε, θεσμικών οργάνων είναι σαφής. Η δημιουργία μιας εσωτερικής αγοράς ενέργειας, βιώσιμη χρήση των εναλλακτικών πηγών ενέργειας, ανταγωνιστικότητα και ασφάλεια στη διαχείριση και στην ε, ανεφοδιασμό της ενέργειας. Αυτή είναι η βασική στόχη της ενεργειακής πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως έχει καθοριστεί από τα θεσμικά όργανα. Είναι προφανές πως οι στόχοι αυτοί για την ενεργειακή πολιτική δεν μπορούν να επιτευχθούν άνευ ορισμένων υποδομών που θα πρέπει ακριβώς να προσαρμοστούν σε αυτό το ενεργειακό πρότυπο. Το ενεργειακό πρότυπο που έχουν ε, θεσπίσει και υπερασπίζονται οι ευρωπαϊκοί θεσμοί. Από αυτό απορρέει η ανάγκη αυτή τη έκθεση που έχει σχέση με τι υποδομέ και με τι προτεραιότητε σε σχέση με τι υποδομέ. Επίσης ε, θα πρέπει να βασιστούμε στην κατάλληλη νομοθετική στήριξη γιατί η συνθήκη της Λισαβόνας μας ορίζει ως ε, συμμετέχοντες στη διαδικασία καθορισμού αυτής της ενεργειακή πολιτικής και Κατά τέταρτο λόγο θα πρέπει να θυμίσουμε ότι με τον καθορισμό των ενεργειακών προτεραιοτήτων και των ε, προτεραιοτήτων σχετικά με τις υποδομές ε, ξεκινάμε σε ένα νέο δρόμο. Ένα δρόμο όμως που πίσω του έχει πολύ παράδοση. Δηλαδή προερχόμαστε, έχουμε μια βάση νομοθετική σε θέματα ενέργειας, την οποία θα πρέπει να εφαρμόσουμε και όχι να ξεχάσουμε. Είναι ο πειρασμός των ευρωπαϊκών θεσμών να προσεγγίζουν το τάδε ή δίνα θέμα και να τίνουν να ξεχνούν τα προηγούμενα βήματα. Ενώ εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να θυμόμαστε τα πράγματα που έχουμε ήδη επιτύχει και που ε, στο θέμα της ενεργικής πολιτικής είναι πολύ σημαντικά. Μιλάμε για σημαντικά νομοθετικά μέτρα όπως το τρίτο πακέτο της εσωτερικής αγοράς, η ρύθμιση της ε, ασφάλειας, ε, για, της ενεργειακής ασφάλειας και επίσης να επιστήσω ιδιαίτερα στην προσοχή σας στο γεγονός ότι η πολιτική για τις νέες ενεργειακές υποδομές όπως και η ενεργειακή πολιτική εν γέννη θα πρέπει να είναι σε συνοχή με τις υπόλοιπες πολιτικές που επιδιώκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως αποτελεί τμήμα ενός συνόλου. Ενός συνόλου που στόχο έχει οι Ευρωπαίοι να ζουν καλύτερα και να επιτύχει τους στόχους που θέτει η συνθήκη της Λισαβόνας. Άρα λοιπόν θα πρέπει να αναζητήσουμε συνοχή ανάμεσα στα όσα κάνουμε εδώ με τους μηχανισμούς για παράδειγμα προστασίας του περιβάλλοντος, ε, καταπολέμησης των κλιματικών αλλαγών, πολιτικής μεταφορών, όλα αυτά είναι ένα σύνολο. Και ένα τμήμα αυτού του συνόλου είναι η ενεργειακή πολιτική και εντό τη ενεργειακή πολιτική με τη σειρά τη και η πολιτική υποδομών με τι προτεραιότητέ τη. Αυτές οι προτεραιότητες και αυτές οι πολιτικές ενεργειακές ήδη υπάρχουν ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και χρόνια. Μόνο που αυτή την περίοδο θέλουμε να ξεπεράσουμε ένα πρότυπο προγραμματισμού, ένα πρόγραμμα προγραμματισμού το οποίο έχει αποτύχει. Αυτό είναι η αποτυχία Να ξεπεράσουμε αυτή την σημερινή συγκυρία όπως έχει μέχρι σήμερα. Για να δούμε τώρα πώς θα συνεχίσουμε όσον αφορά αυτή τη νέα πολιτική θα θέλουμε να επιδιώξουμε, να πετύχουμε κάποιους ξεκάθαρους στόχους, να υπάρξει η, διανομή, των μοίρα Μετρική ενέργεια με δίκτυα και επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω το πόσο σημαντικό είναι αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε. Δηλαδή θέλουμε να έχουμε αυτές τις ευφυείς πόλεις, το οποίο πάνε να πει πόλεις ε, οι οποίες να είναι αφοσιωμένε στην προστασία του περιβάλλοντος, να είναι δεσμευμένε ή στο να φροντίζουν για να υπάρχει οικονόμηση ενέργειας και άρα να υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί για την κατανάλωση ενέργειας του πολίτη. Πάρα πολύ σημαντική είναι αυτή η προοπτική και αυτό θα εμπλέξει τις ε, αρχές παντός επίπεδου, παντός είδου ή στην Ευρώπη. Ε, δημοτικές αρχές, ε, ε, οι δήμαρχοι, το δημαρχία. Δηλαδή μιλάμε για κάποιους οι οποίοι πολλές φορές ε, τους, τους, τους ξεχνάνε οι Βρυξέλλες. Επίσης θα θέλουμε να υπάρχει αποτελεσματική ε, κατανομή και διανομή της ενέργειας και του φυσικού αερίου. Αλλά θέλω τώρα να σταθώ όσον αφορά αυτή την, την καινούργια προσπάθεια τα εξή δύο πρώτα πρώτα να μειώσουμε την εξάρτησή μας από το εξωτερικό και δεύτερον θέλουμε να τελειώσουν αυτού του είδους οι ενεργειακές νησίδες που υπάρχουν. Είναι αυτές οι δύο οι, αυτές οι, δύο, οι, έννοιες που πρέπει να τις φροντίσουμε όσον αφορά την ενέργεια. Οπότε γι' αυτό θέλουμε τώρα να θέσουμε σε κινητοποίηση αυτό που ονομάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενεργειακούς διαδρόμους. Κατά δεύτερο λόγο ε, ε, έχουμε ε, αυτά τα ονομαζόμενα έργα ή προγράμματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό τώρα πρέπει να κάνουμε να καθορίσουμε κάποια κριτήρια. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει μια ιεραρχία όσον αφορά τα κριτήρια την ώρα που θα έρθει για να μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε τι θα γίνει με αυτά τα ε, προγράμματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Οπότε θα πρέπει συνεργούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάτσουμε και να χτενίσουμε αυτά τα κριτήρια, να είμαστε ακριβείς και να μπορέσουμε να προοδεύσουμε όσον αφορά την περιχαράκωση αυτών των ε, κριτηρίων διότι πρόκειται για κάτι που θα είναι πάρα πολύ θετικό για το να πετύχουμε αυτά που θέλουμε στους αμέσους μήνες. Πρόκειται επομένω για κάποια κριτήρια τα οποία είναι η εξοικονόμηση ενέργειας, ε, η χρήση, η λελογισμένη των υποδομών που υπάρχουν και γι' αυτό και εγώ τώρα ζητώ από τα μέλη της Επιτροπής, τους συναδέλφους για όλα αυτά τα οποία έχουμε κάνει από κοινού να με βοηθήσουν λέγω να κάνουμε και άλλα και η Επιτροπή να μπορέσει να κάνει περισσότερα όσον αφορά την υπόθεση αυτή. Ένα πρόβλημα τώρα το οποίο μας ε, προβληματίζει πάρα πολύ τώρα που ήρθε η ώρα να καθορίσουμε τις προτεραιότητες είναι το πρόβλημα των ε, εγκρίσεων, αδειών, ε, αδειοδοτήσεων κλπ. όσον αφορά και τους 27 για την ενεργειακή πολιτική. Είναι πολύπλοκο αυτό γιατί έχουμε να κάνουμε ένα σωρό εθνικές νομοθεσίες και σε κάθε χώρα ε, πολλές φορές υπάρχει εθνική και όχι κοινωτική αρμοδιότητα. Όμως εμείς θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθεια, διότι πρόκειται εδώ για ένα κομβικό κεντρικό πρόβλημα, μια που ε, πολλές φορές ε, τα προγράμματα αυτά τρέχουν για παραπάνω από όσο προβλέπετε, πάμε για δεκαετίες ή παραπάνω και εδώ εμπλέκονται διάφορες αρχές, κρατικές, περιφερειακές και εδώ μπλέκεται το θέμα όσον αφορά τι αδειοδοτήσει, τι συγκρίσεις και θα πρέπει για όλα αυτά οι προθεσμίε να είναι ξεκάθαρες. Επομένω, τώρα μιλούμε για κοινοτική νομοθεσία και εναρμόνιση για όλα αυτά για να δούμε τι γίνεται και πώ μπορεί η κοινοτική νομοθεσία να παρέμβει, να προσπαθήσει να εναρμονίσει τα των εθνικών νομοθεσιών τα πιο σημαντικά. Δηλαδή πρώτα-πρώτα τις ε, προθεσμίες καταληκτικές ημερομηνίε για αυτά τα προγράμματα που λέμε επίσης να δούμε τι θα γίνει για την διοικητική σιωπή δηλαδή πολλές φορές όταν έχουν αρμοδιότητα αδρανούν οι, αρχές οπότε να δούμε τι θα γίνει με αυτό ε, λέμε εδώ πέρα για αυτό το ενιαίο μοναδικό παράθυρο ήγισε. Αυτή τη θηρίδα. Γιατί μιλούμε τώρα για πολλές φορές για χρήσεις, για συνοήσεις διασυνοριακές για αυτή την ενιαία θηρίδα. Οπότε έχουμε τέτοια προγράμματα που τρέχουν σε περισσότερο από ένα κράτη οπότε θα πρέπει να κάτσουμε και να επεξεργαστούμε περισσότερο το, το θέμα, <laughs> πιο ενδέλεχος. Και επίσης να δούμε τι θα γίνει με την επικουρικότητα. Είναι πάρα πολύ βασική αρχή όσον αφορά την ε, κοινοτική δικαϊκή τάξη και επίσης θα πρέπει να φροντίσουν να υπάρχουν εγγυήσεις για να εμπλέξουμε στα προγράμματα αυτά τον κόσμο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ο κόσμος να αισθάνεται ότι είναι δικά του αυτά τα προγράμματα και τα έργα. Οι φορείς των πολιτών μπορούν να κάνουν πάρα πολλά. Το έχει δείξει αυτό η εμπειρία μας. Ότι ή μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ ή μπορούν να το υπονομεύσουν τελείως το, το έργο ή το πρόγραμμα. Άρα θα πρέπει από τη γέννηση, από την αρχή, από την πρώτη μέρα που τρέχει ένα πρόγραμμα να εμπλέκεται ο κόσμος και να ξέρουμε κάθε φορά τι εναλλακτικέ τεχνικές υπάρχουν, να τα ξέρει και ο κόσμος και αυτό γιατί νομίζω ότι ε, ε, έχουμε προχωρήσει όσον αυτό και τελικά δεν είναι αλήθεια ότι είναι αποξενωμένος ο κόσμος διότι έχει βοηθήσει η, η νομοθεσία υπάρχουν ένα σωρό τεχνικές, θετικές όμως πρέπει να επιμείνουμε περισσότερο το σημείο τώρα για τη χρηματοδότηση για τη χρηματοδότηση αυτό το οποίο λέω στην έκθεση είναι ότι θα πρέπει να είναι του ιδιωτικού τομέα η χρηματοδότηση να πληρώνει δηλαδή όποιος καταναλώνει. Άρα ο τομέα τομέας όμως δεν αποκλείουμε να υπάρχει και συμμετοχή του, δημο, του δημοσίου τομέα μια που από εμπορική, αλλά κυρίω γιατί υπάρχει ενδιαφέρον ευρωπαϊκό ενδιαφέρον για το κράτος. Θα πρέπει τώρα η Επιτροπή αλλά και εμείς να προσπαθήσουμε να δούμε περισσότερο το τι προβλήματα δημιουργούν αυτά τα διασυνοριακά προγράμματα. Ποιος πληρώνει, πώς γίνεται η κατανομή της συμμετοχής στο κόστος και πέρα από τα προβλήματα αυτά της χρηματοδότησης να δούμε τι ζητούν όλοι όσοι εμπλέκονται στην υπόθεση ενέργεια και άρα χρειάζεται κάποιο ρυθμιστικό πλαίσιο. Το χειρότερο από όλα για τα ενεργειακά προγράμματα, βέβαια ισχύει για, όλα, είναι το να έχουμε αλλαγές, να έχουμε πισωγυρίσματα όσον αφορά την νομοθεσία, γιατί αυτό είναι τραγικό, είναι θανάσιμο για αυτούς οι οποίοι συμμετέχουν και τρέχουν τα προγράμματα. Επομένως να υπάρχει ένα σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο. Αυτό πρόκειται να λύσει για τα προβλήματα της χρηματοδότησης. Για όλα αυτά έχω αποφανθεί ή στο έγγραφο το οποίο σας έχω υποβάλει ως συγητής και βεβαίως ε, να συμπληρώσω την ενημέρωσή σας να, να τα να, να, να, να χτενίσω, να διορθώσω αυτά τα οποία είπα ανάλογα με το τι τυχόν έχετε να προτείνετε. Επίσης πρέπει να σας πω ότι εδώ ε, υπήρξε συνεργασία αγαστή, πολύ καλή με όλους τους ε, συναδέλφους και έχουμε επομένω τώρα μια ε, συνεργασία πάρα πολύ φιλική, πάρα πολύ αποδοτική και ελπίζω ότι μέχρι ότου ολοκληρωθεί η δουλειά μου ότι όλα θα πάνε το ίδιο καλά. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Πρέπει να μην ξεχνάμε και το ρολόι. Okay. Θα σας ευγνώμουν λοιπόν αν είσαστε κάπως σύντομοι όταν ζητάτε το λόγο. Θα τρέχει το ρολόι εδώ και έχουμε ακόμα και τη... αυτούς που έχουν ζητήσει το λόγο από την περασμένη φορά. Θα πάρουν το λόγο αυτοί που έχουν ζητήσει το λόγο την περασμένη φορά γιατί τους το είχαμε υποσχεθεί και μετά οι σκιώδεις Καταρχήν η κυρία Κουλάσκα Κουλάσκα-Βομπίνσκα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ενδιαφέρον που θυμόσαστε ποιοι είχαν ζητήσει το λόγο την περισμένη φορά. Καταπληκτικό. Ένα από τα πράγματα που θα πρέπει να σκεφτούμε στην έκθεσή μας είναι κάτι που ανέφερε και ο συγητής και θα αναφέρουν και άλλοι συγητές, δηλαδή τα κριτήρια για την επιλογή των διαφορών σχεδίων. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να έχουμε κατά νου. Και θα πρέπει να αποδώσουμε ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός ότι ε, κάθε σχέδιο που θα βοηθήσει θα πρέπει να τηρεί τουλάχιστον δύο κριτήρια. Γιατί υπάρχουν διάφορα σχέδια στα οποία πληρούνται δύο Λοιπόν, θα πρέπει να επιλέξουμε εκείνα που χρειάζονται 2 εις 3. Θα πρέπει παραδείγματο χάρη να αποδώσουμε προσοχή και σε έναν ορισμό ευρωπαϊκού σχεδίου. Η Κομισιόν είπε παραδείγματο χάρη ότι το Nord Stream είναι ευρωπαϊκό σχέδιο αλλά δεν θα χρειαστεί ε, ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Κατά πόσο λοιπόν είναι ευρωπαϊκό, γιατί αν δεν κάνω λάθος ο Επίτροπος ανέφερε ότι θα ε, έχουμε μια ασφάλεια τροφοδότησης. Ένα κριτήριο είναι αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να εργαστούμε πάνω στον ορισμό του τι είναι το ευρωπαϊκό σχέδιο και τι θα πρέπει να πληρούνται με αυτό. Κάτι άλλο που θα πρέπει να σκεφτούμε είναι η χρηματοδότηση. Και εδώ η άποψή μου είναι ότι δεν θα πρέπει να εφαρμόσουμε νέα μέσα για η δημιουργία νέων μέσων χρειάζεται χρόνο, αξιολόγηση, χρειάζεται αρκετός χρόνος δηλαδή για να γίνει κάτι τέτοιο και θα πρέπει να εργαστούμε προσεκτικά στα σχέδια υποδομής και τρίτον όταν συζητάμε στα πανευρωπαϊκά δίκτυα συνήθως αναφέρουμε τη δημιουργία νέων διασυνδέσεων και νέων κατευθύνσεων. Σημαντικό αυτό, αλλά το ευρωπαϊκό σύστημα πρέπει να είναι συνεπές, θα πρέπει να έχουμε κατά νου και τον ε, εξυγχρονισμό με εκείνα τα δίκτυα που έχουν φτάσει στο τέλος της ζωής τους και δεν θα είναι πια λειτουργικά και τμήμα του ευρωπαϊκού δικτύου. Εν κατακλείδη, Πρόεδρε, θεωρώ, είναι καλό να σκεφτόμαστε αυτά τα σχέδια στην Βόρειο Θάλασσα και να μην ξεχνάμε και την Αφρική, αλλά να θυμάμαι και εκείνες τις χώρες που έχουν κάποια δίκτυα, ηλεκτρικά δίκτυα δηλαδή, που δεν είναι ακόμα επαρκώς ανεπτυγμένα. Υπάρχουν τεράστιοι τομείς στην Ευρώπη όπου λείπουν οι διασυνδέσεις. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Βίταλ παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αναμφίβολα έχουμε εδώ στα χέρια μας μια έκθεση πάρα πολύ σημαντική διότι η Επιτροπή μας και γενικότερα τα θεσμικά όργανα εδώ και 10 χρόνια προσπαθούμε να δούμε τι θα κάνουμε για την ε, ενιαία αγορά που θέλουμε να είναι απελευθερωμένη ε, και μιλούμε για την αγορά της ενέργειας ε, και να είναι μια αγορά πανευρωπαϊκών διαστάσεων που να μπορεί να είναι ανταγωνιστική, να μπορεί να βοηθήσει να βελτιώνεται το βιωτικό επίπεδο του κόσμου και νομοθετούμε και ξανανομοθετούμε πρόσφατα και ε, είμαστε φιλόδοξοι στις προσπάθειές μας οπότε και η σημερινή έκθεση ε, έρχεται να άρει ένα κενό το οποίο υπήρχε διότι εάν δεν ε, υλοποιηθεί αυτό το οποίο επιδιώκουμε όλα τα υπόλοιπα γίνονται μάταια. θα πρέπει επομένως να δούμε τι γίνεται για όλε αυτές τις δέσμες μέτρων που έχουμε περάσει όσον αφορά την εσωτερική αγορά ενέργειας. Έχουμε κάνει ένα σωρό πλάνα και σχέδια για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί σε αυτή την ενεργειακή αγορά. Όμως αν δεν υπάρχει μια υποδομή, αν δεν υπάρχει κάτι απτό, χειροπιαστό που να βοηθάει ε, τα υπόλοιπα, τότε, τότε όλα είναι επεαπτερόεντα αυτά τα οποία κάναμε. Και γι' αυτό σας λέω ότι τώρα φτάσαμε σε ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο της διαδρομής για να πετύχουμε το στόχο μας που είναι η ολοκλήρωση αυτής της αγοράς ενέργειας και όλα τα οποία είπε ο εισηγητής μου αρέσαν εμένα επομένως και όσον αφορά το περιεχόμενο των όσων είπε αλλά και το ότι επέδειξε μια τέτοια διάθεση που μου φαίνεται ότι είναι πραγματική, ειλικρινής να δουλέψουμε σαν μια ομάδα και να συνεργαστεί με τους σκιώδες εισηγητές. Με την ευκαιρία τώρα πρόεδρε θα πρέπει να δούμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας έδωσε μια καλή αφετηρία που είναι αυτό το έγγραφο, αυτό το δεν ισχύει πάντοτε. Πολλές φορές έρχεται κάτι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το οποίο απέχει πόρα από αυτό το οποίο εμείς πρεσβεύουμε. Όμως εν προκειμένου ε, σε εμά και στο Συμβούλιο ε, κατέβασε κάποιες προτάσεις που νομίζω ότι πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση που αποτελούν τα αναγκαία συστατικά για να μπορέσουμε να εργαστούμε αποδοτικά. Να δούμε τώρα τα πιο συγκεκριμένα σημεία. Αναφέρθηκε ο συγητής σε κάποιες διοικητικές διαδικασίες και συγκεκριμένα σε εγκρίσεις και αδειοδοτήσει δύσκολα θέματα αυτά, ιδίω όταν έχουμε προγράμματα που αφορούν πάνω από ένα κράτος μέλος διασυνοριακά και επομένω. όπως ελέγξτε θα πρέπει ενωσιακά να υπάρξει κάποια ρύθμιση για απλούστευση, για κινητοποίηση όμως αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο και πρέπει και να τηρείται πάντοτε και η επικουρικότητα όμως έχουμε εργαλεία Έχουμε εργαλεία που μας επιτρέπουν να επιτύχουμε βήματα πρόοδου, να τα χρησιμοποιήσουμε και να αξιοποιήσουμε αυτή την έκθεση. Τώρα υπάρχουν όμως και κάποιες άλλες περιπτώσεις ε, κατά τις οποίες η δυσκολία αναδύεται από το ότι δεν υπάρχουν κίνητα, δεν υπάρχει ενδιαφέρον για τους επενδυτές για κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα ή έργο. Οπότε, είναι προκειμένου, αυτό που θα πρέπει να φροντίσουμε να κάνουμε είναι οι κυβερνήσεις με ε, κάποιο είδους κατάλληλη τιμολογιακή πολιτική η φορολογική πολιτική να μην αποθαρρύνουν τους ενδυνάμει επενδυτές γιατί αλλιώς δεν θα ενδιαφέρονται και άρα θα κολλήσει το πρόγραμμα. Δεν είναι δυνατόν οι τιμή ενέργειας να είναι κάτω από το κόστος της παραγωγής ενέργεια αλλά και της ε, διανομή τη. Αυτό νομίζω ότι είναι προφανέ και νομίζω ότι ο βρίσκει σύμφωνο. Επομένω, όταν έχουμε κάποιο πρόγραμμα το οποίο είναι ελκυστικό από πλευρά οικονομική, θα πρέπει τότε να μην το φρενάρουμε με νομοθεσίες, με ρυθμιστικά μέτρα τα οποία αντιβαίνουν στην ε, οικονομική πραγματικότητα. Οπότε θα πρέπει να δούμε πώς θα έχουμε μια εύστοχη πολιτική, μια πετυχημένη πολιτική για υποδομές, για ενέργεια. Ε, θα πρέπει να κάτσουμε και να συμπληρώσουμε την ήδη κοιμή νομοθεσία. Έχουμε τώρα την τρίτη δέσμη μέτρων για την ιστορική αγορά ενέργειας και επίσης έχουμε και τον κανονισμό για την ε, ασφαλή προμήθεια φυσικού αερίου. Όλα αυτά είναι απαραίτητα συστατικά για την πολιτική των, ε, ε, των μέτρων ε, των, των έργων υποδομής και επομένως θα πρέπει να δούμε πώς θα συμπλώσουμε την κείμενη νομοθεσία όπως είπαμε και σε περίπτωση που υπάρχει καθυστέρηση θα πρέπει να δούμε πώς θα έχουμε κάποιο είδους θεμητή επιτρεπόμενη αναγκαστική εκτέλεση του υπήν για εκεί που υπάρχουν οι καθυστερήσει. Να δούμε τώρα ε, σε ποια έργα υποδομή θεωρούμε ότι έχουν ε, την υψίστη προτεραιότητα για την παροχή της ενέργειας είναι πάρα πολύ σημαντικά τα έργα υποδομής και έτσι να μπορέσουμε και να καταπολεμήσουμε την αλλαγή του κλίματος οπότε πολλές φορές πρέπει να υπάρχει ε, κρατική συμβολή οικονομική και έτσι τα προγράμματα να είναι ε, να είναι ελκυστικά για τις αγορές. Αυτό μπορεί να γίνει τώρα με δύο τρόπους. Ή μπορεί κάποιος απευθείας να έχει ε, αυτή τη λύση της λίστας ή θα μπορούσε κανείς να έχει καθορίσει εκ των προτέρων κάποια κριτήρια η προσωπική μου γνώμη, αλλά νομίζω και του συγκεκριτή από ό,τι καταλαβαίνω, είναι το ότι το πιο σωστό είναι ευθύ εξ αρχή να μου καθοριστεί κάποια κριτήρια επί των οποίων οι πάντε να συμφωνούν. Για παράδειγμα, ε, κατάργηση των ενεργειακών νησίδων. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε πάνω σε αυτό. Όταν επομένω κάποιο κράτο μέλο εξαρτάται πάρα πολύ από έναν και μόνο ε, πάροχο ενέργειας ε, και έχουμε αντίστοιχα κάποια έργα τα οποία αποσκοπούν στο να άρουν αυτή την αποκλειστικότητα. Ε, συμφωνούμε όλοι ότι αυτό είναι ένα σωστό κριτήριο. Και για τον ίδιο λόγο σας λέω ότι χρειάζονται κάποιες υποδομές, που να βοηθούν την ε, περιφερειακή συνεργασία. Και επομένως, ε, όταν έχει να αντιμετωπίσουμε πιο συγκεκριμένα ζητήματα, τότε ε, θα έχουμε ήδη μειώσει στο μέγιστο βαθμό τα σημεία προστριβής. Γι' αυτό σας λέω, Πρόεδρε, έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Ξεκινήσαμε όμως καλά. Και βέβαια και ο καθηγητής Σώσα Βάγνερ μπορεί να υπολογίζει στην δική μας ε, συνεργασία και βοήθεια ούτως ώστε να έχει αίσιο πέρας αυτή η υπόθεση. Σας ευχαριστώ και εγώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ο χρόνος που μιλάει ο κανένας θα αναγραφεί για τον καθένα μπροστά σας. Θα το δείτε. Και αν δεν μπορέσουμε να περικόψουμε, δεν θα μπορέσουν να μιλήσουν όλοι. Θα ήθελα να προτείνω λοιπόν ο καθένας δύο λεπτά. Κάριντς, επόμενος μιλητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ με εκείνους που μιλήσανε πριν από μένα. Διάβασα προσεκτικά το έγγραφο εργασία που υπέβαλε ο εισηγητής και θα ήθελα να αφαιρθώ μόνο σε ένα θέμα. Και αυτό είναι κάτι στο οποίο ανέφερε και ο κύριος Βίδαλ Είναι σαφές ότι για να πετύχουμε την υποδομή είναι το πιο σημαντικό, γιατί αν δεν έχουμε μια κοινή υποδομή για την ενέργεια, δεν θα πετύχουμε τίποτα. Και αυτό θα είναι καλός στόχος για τον Ευρωπαίο καταναλωτή. Η δυσκολία είναι ότι ορισμένα από τα σχέδια μπορούν εμπορικά να επιβιώσουν και δεν θα είναι δύσκολο να ε, προσελκύσουν χρηματοδότηση. Θα υπάρχουν όμως και άλλα σχέδια τα οποία δεν θα είναι αμέσως οικονομικά επιβιώσιμα και θα χρειάζονται δημόσιο χρήμα. Το θέμα λοιπόν είναι ποια θα είναι αυτά τα σχέδια, πώς θα το αποφασίσουμε και ποια θα είναι εκτός του δημοσίου χρήματος δηλαδή. Γιατί ορισμένοι ενδιαφέρονται βέβαια να έχουν κάποια δημόσια χρήματα για να μειώσουν το κόστος της επένδυσης. Είναι λογικό αυτό. Για να μην λοιπόν κατακαιρματίσουμε το λίγο δημόσιο χρέμα που θα διατίθεται, είναι σωστό να ακολουθήσουμε την άγουσα του ο εισηγητή. Και στη σελίδα 6 λέει ότι για να μην ε, κατασπαρθούν τα λίγα οικονομικά βοηθήματα που θα υπάρχουν, θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια πιο λογική μεθοδολογία. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν λογικό. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να έχουμε ένα κατάλογο των σχεδίων, αλλά να έχουμε μια μεθοδολογία θα, για το ποια είναι αυτά τα σχέδια που θα χρειαστούν την δημόσια χρηματοδότηση, θα μπορέσουμε νομίζω να βοηθηθούμε. Είναι αυτή μια από τι κυρίες μα προκλήσει, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Μαντουέλ έχει το λόγο. <coughs> gracias, presidente, yo también felicitar al ponente por su trabajo y decir que básicamente. Ε, ευχαριστούμε κύριε Σιγητά για αυτά που κάνατε. Συμφωνώ με τα όσα είπατε. Όμως θα ήθελα να σας πω κάποιες σκέψεις μου. Το είπατε, το είπε ο Βιδάλ Κουάδρος, θα πρέπει να καταργηθούν οι νησίδες οι ενεργειακές. Και γι' αυτό και εγώ θέλω να σας πω κάτι συγκεκριμένο. Θα πρέπει να το ξαναπείτε στην έκθεση το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να φτάσει το 10% όσον αφορά τη δυνατότητα διασύνδεσης που αποφασίστηκε στο Συμβούλιο της Βαρκελόνης. Γιατί θα πρέπει να συνεχίσουμε επειδή έχουμε αυτό το στόχο, όπως και τους άλλους στόχους για, τη, για τα ανανεώσιμα, για το 2020 κλπ. Είναι σαφές ότι η ανάπτυξη των υποδομών ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος δεν είναι δυνατόν να εξαρτάται μόνο από την βούληση των κρατών μελών. Το επιπημένω σε αυτό θα πρέπει να υπάρχουν και κριτήρια ε, εμπορικά. Είναι πάρα πολύ χρήσιμα αυτά τα αναπτυξιακά σχέδια και τα είπαμε από τον Ιούνιο. Ε, είπαμε ότι χρειάζεται συνεργασία, συντονισμός, ε, δεν υπάρχει ευρωπαϊκό όραμα το οποίο να είναι συνολικό και σφαιρικό τα ξέρετε, ξεκαθαρίστηκαν, δεν το ξαναλέω τώρα για τη χρηματοδότηση. Έχουμε ως αφετηρία το ότι η χρηματοδότηση των υποδομών θα πρέπει να είναι σύντονο να υπόκειται στα κριτήρια της αγοράς, του είπε οπότε όμως κάθεται και λέει η Κομισιόν ότι χρειάζονται 100 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό πάρα πολύ δύσκολο θα γίνει. Όμως ε, είναι απαραίτητο, όπως είπε και ο εισηγητής, να αυξηθούν οι, οι πόροι στον προϋπολογισμό για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε εκείνες τις υποδομές βρίσκοντας την ε, απαραίτητη χρηματοδότηση τέλος ε, για τους καταναλωτές θέλω κάτι να πω συχνά ακούμε τα επιχειρήματα ότι δεν μπορούμε να επενδύσουμε σε υποδομές διότι κατά τον τρόπο θα οδηγηθούμε σε αύξηση της τιμής της ενέργειας. Όμως όλοι γνωρίζουμε το κόστος των υποδομών είναι το ελάχιστο κομματάκι της διαμορφούμενης τιμής ενέργειας. Ας πούμε για τη χώρα μου που ξέρω, για το φυσικό αέριο είναι κάτω από το 10% της διαμορφούμενης τιμής το κόστος της, ε, της υποδομής. Γιατί έτσι έχουμε πιο ολοκληρωμένε αγορές, περισσότερη διασύνδεση και έχουμε και έτσι και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Ε, και τελικά και οι τιμές διαμορφώνονται σε εφικτά επίπεδα και άρα οι υποδομές τελικά είναι εις όφελος των καταναλωτών. Επαναλαμβάνω Πρόεδρε ότι στενά θα συνεργαστώ με τον εισηγητή και επίσης τα συγχαρητήριά μου για το έγγραφό του. Για ενημέρωσή σας έχουν ακόμα 10 που έχουν ζητήσει το λόγο και πριν από τις 10 έχουμε και άλλο ένα θέμα κατά βάση. Συνάδελφος το έχει το λόγο. Monsieur le Président. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Προφανώς να υπογραμμίσω και το λέω με ειλικρίνεια και να συγχαρώ τον εισηγητή για την εργασία του και για το πνεύμα συνεργασίας που έχει δείξει. Ε, έχω να πω τα εξής. Όταν ε, ε, μιλάμε για την, ε, τις υποδομές ε, μέχρι το, με τον ορίζοντα του 2015. Θα, δεν θα ήταν ρεαλιστικό να μιλάμε για ενέργεια αν οι υποδομές που υπάρχουν ακόμα σε εκείνη την περίοδο δεν αντιστοιχούν σε αυτές τις προβλέψεις που κάνουμε για το 2050. Επίσης θα πρέπει να δοθεί μια, ένα είδος ε, ιεραρχίας, ε, ιεράρχησης μάλλον των υποδομών. Έχουμε κάνει ήδη αυτή τη συζήτηση και ο εισηγητής διοργάνωσε μια συνεδρίαση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πρότυπο το ίδιο το οποίο διέπει την εργασία της Επιτροπής. Γνωρίζουμε πως δυνητικά πρόκειται και 140 δις ευρώ επενδύσεις, αλλά ότι αν υπάρχουν και άλλα ενεργειακά πρότυπα, που λένε ότι αν επενδύαμε ε, ε, σοβαρά στις εξοικονομίες ενέργειας ε, θα φτάναμε στα 70 δις θα κάναμε μεγάλες οικονομίες. Δηλαδή υπάρχει βασική πρόκληση λοιπόν όσον αφορά τα ευρώ που επενδύουμε αλλά και το ενεργειακό πρότυπο. Και εγώ θα πρότεινα Προέδρε η Επιτροπή μας να κάνει μια επίσημη, ένα επίσημο αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε σε όλη την, το εγχείρημα του Energy Roadmap που αναπτύσσεται να γίνει μια συζήτηση σε σχέση με το ποιο πρότυπο θα χρησιμοποιήσει η Κομισιόν. Δεν είναι φυσιολογικό για τόσο σοβαρά θέματα η Κομισιόν Κομισιόν να προσκολάται σε ένα μόνο πρότυπο και να μην υπάρχει μια αντίθετη γνώμη για το πρότυπο που χρησιμοποιείται. Τρίτο σημείο, το θέμα των προτεραιοτήτων όσον αφορά τις υποδομές που θα πρέπει να στηριχτούν. Φυσικά θα πρέπει να τεθούν προτεραιότητες ε, όσον αφορά τους διαδρόμους αλλά και ανάμεσα και στους διαδρόμους προτεραιότητας. Εμείς θεωρούμε πως τρεις είναι οι βασικές προτεραιότητες που αντιστοιχούν σε τρεις επίγουσες καταστάσεις. Πρώτον, το υπερδίκτυο με το δίκτυο της Βόρειας Θάλασσας. Θα πρέπει να συνδεθεί κάθε δυνατότητα για σύνδεση της Βόρειας Θάλασσας με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο. Και έπειτα ο διάδρομος Ανατολή Δύση για το φυσικό αέριο με διπλή ροή είναι πολύ σημαντικό για την αλληλεγγύη Ανατολή Δύση και έπειτα το θέμα των απομονωμένων περιοχών. Και αυτό ήδη Η διαδικασία αδειοδότησης για τις νέες υποδομές θέλουμε να πάνε γρήγορα τα πράγματα φυσικά, αλλά ένα πρόγραμμα το οποίο δεν έχει συζητηθεί με του τοπικούς πληθυσμούς είναι ένα, ένα σχέδιο το οποίο μπορεί να καθυστερήσει και να ε, χρονοτριβήσει. Πρέπει δηλαδή να γίνουν διαβουλεύσει σε τοπικό επίπεδο. Και ένα πέμπτο σημείο. Σε αυτό το έγγραφο δεν μιλάμε για Ε, την ε, διαρροή άνθρακα μπορεί να υπάρξει κάτι τέτοιο ε, ειδικά όσον αφορά τις ενεργειακές δομές εκτός της Ένωσης και έπειτα στην έκθεση το θέμα το φυσικό αέριο από σχιστόλιθο το χρησιμοποιούν στη Βόρεια Αμερική, γιατί δεν μπορούμε να βάλουμε και εμείς αυτό το θέμα εδώ. Ε, είναι πάρα πολύ τοξικό, είναι πραγματικά φρικτό από την άποψη του περιβάλλοντος και της διαχείρισης του περιβάλλοντος. Ε, το δυναμικό βιώσιμης χρήσης του φυσικού αερίου, όπως χιστόλιθο, είναι μηδενικό. Ε, θα ήθελα λοιπόν το θέμα αυτό να μην συζητηθεί καν, γιατί δεν είναι σοβαρό θέμα. Λοιπόν, δεν θα μπορέσω να δώσω το λόγο σε όλους τους συνάδελφους να συνεχίσουμε έτσι. Συνάδελφος Παλαιάν. Uh, ευχαριστώ. Θα τα πω γλυκόρα παρόλο που είμαι και η εισηγήτρια για τις φιλελεύθερους. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστώ τον εισηγητή για την τόσο χρήσιμη και κατανοητή εργασία που έκανε στο έγγραφό του και επίσης θα ήθελα να πω ότι ακτιμώ την φιλοδοξιστάση τη της Κομισιόν στη δέσμη αυτό. Είναι πολύ είναι πολύ σημαντικό αυτό το βήμα. Όταν μιλάμε τώρα για τις επενδύσεις στις υποδομές, θα πρέπει να τονίσουμε στο 2050 και για να ενθαρρύνουμε την Κομισιό να υπάρχει σωστή ε, συνοχή με το χρονοδιάγραμμα για το 2050 και τους στόχους για το 2020. Δεύτερον, θα ήθελα να σας πω ότι στο οικονομικό πλαίσιο της σήμερα θα πρέπει να ξεχνάμε ότι χρειαζόμαστε όλα τα μείγματα ενέργειας που μπορούμε και να μην αποκλείουμε κάποιες πηγές ενέργειας ως ηθικά απαράδεκτες. Κατόπιν, όσον αφορά το μέγεθος των σχεδίων, αντί να ρίχνουμε τεράστια ποσά της Ευρώπης σε τεράστια έργα, θα πρέπει να εξτάσουμε ίσως μικρά και πιο αποτελεσματικά σχέδια, που θα μπορέσουν πραγματικά να προσφέρουν γλίγορα μια προστιθέμενη αξία. Συμφερίζω με τις απόψεις εκείνων που είπαν ότι χρειαζόμαστε πολύ ξεκάθαρα κριτήρια και ξεκάθαρη ιεράρχηση μεταξύ των διαφόρων σχεδίων που θα εξετάζουμε. Και όσον αφορά την οικονομική πλευρά, έχω να πω ότι χαιρετίζω την προσέγγιση της Κομισιόν για χρηματοδότηση βασιζόμενη στην αγορά από την άλλη μεριά νομίζω ότι χρειαζόμαστε νέα χρηματοδοτικά μέτρα να ξετάσουμε το θέμα χρεογράφων και εταιρική σχέση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να προχωρήσουμε στον τομέα ιδίω των υποδομών. Τελευταίο σημείο που θα ήθελα να παρουσιάσω, όπως και άλλοι ομιλητές, θα ήθελα να πω ότι και για μας είναι σημαντικό να υπάρχουν πιο φιλόδοξα ε, μέτρα ιδίως για τα διαμεθορικά σχέδια αυτά πρόεδρε θα, τα υπόλοιπα θα σας τα πω άλλη φορά ευχαριστώ Σιμπάνσκι Dziękuję bardzo. Ja starałem się przeczytać ten komunikat e, raz jeszcze w kontekście... Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Εγώ προσπάθησα να διαβάσω ξανά την ανακοίνωση αυτή δεδομένων των συμπερασμάτων του Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου και μπορούμε σαφώς να δούμε ότι υπάρχουν κάποιες παρατηρήσεις να κάνουμε εδώ. Η ανάπτυξη της, ε, του, του, της, του μείγματος ενέργειας δεν μπορεί μόνο να αντιμετωπιστεί με τη, σε σύνδεση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα πρέπει να συνδυαστεί με τις την εθνική ε, κατάσταση για να χρησιμοποιηθούν και εσωτερικοί πόροι, πηγές ενέργειας. Θα πρέπει δηλαδή να ισχύσουν διάφορα κριτήρια για την ανάπτυξη. Οι διεθνείς συνδέσεις ε, από μόνες τους δεν θα εξασφαλίσουν υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας σε ανεφοδιασμού, ούτε καλύτερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Θα πρέπει αυτά να συνδυαστούν με την ανάπτυξη των εθνικών ε, δικτύων και φυσικά θα είναι κρίσιμη η επιλογή των σωστών προτεραιοτήτων που είναι προς το ευρωπαϊκό συμφέρον. Είμαι βέβαιος πως η αγορά θα μπορέσει να χειριστεί τις επενδύσεις ε, σε κάποιο βαθμό, αλλά ίσως θα μπορούσαμε να, ε, να, να επιδοτήσουμε με ευρωπαϊκά χρήματα μόνο τα προγράμματα που πληρούν κάποια κριτήρια. Αυτό μπορεί να έχει να κάνει με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά ίσως και με την ασφάλεια στην ε, ενέργεια. Και εδώ χρειάζεται διαφοροποίηση. Όχι μόνο για την ε, διαβίβαση της ενέργειας, αλλά και για τις πηγές ενέργειας. Και το στοιχείο που θα πρέπει ιδιαίτερα να προσεχθεί είναι η σύνδεση ανάμεσα στο βορρά και στο νότο από τα πολωνικά, τις πολωνικές δηλαδή αποθήκες φυσικού αερίου στις κροατικές. Χωρίς τέτοιου είδους λύσεις η αγορά δεν θα λειτουργήσει σωστά αποτελεσματικά διότι δεν θα υπάρχουν πρακτικές λύσεις ώστε να λειτουργήσει μια εσωτερική αγορά φυσικού αερίου. Τώρα, για το αέριο από σχιστόλιθο δεν νομίζω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε μόνο τα περιβαλλοντικά ζητήματα εκεί και τις προκαταλήψεις που επικρατούν και δείτε την πυρηνική ενέργεια. Αν είχαμε τέτοια προσέγγιση προς την πυρηνική ενέργεια πριν από κάποια χρόνια, ε, δεν θα είχαμε την ε, πυρηνική ενέργεια σήμερα. Τέτοιο είδους ενεργειακό, μάλλον πιστεύω πως ε, τέτοιο είδους ενεργειακό μείγμα μπορεί να μην χρειάζεται επιδότηση. Όχι, αλλά θα χρειάζεται το κατάλληλο νομικό πλαίσιο ώστε να μην υπάρχει γραφειοκρατία και φραγμή διοικητικού τύπου. Αυτά επιθυμεί ο κλάδος από εμά. Ας μην σκεφτόμαστε λοιπόν μόνο τις, ε, τα cash flows, ε, να σκεφτόμαστε και πώς δεν θα εμποδίσουμε με τις νομοθεσίες μας. Ευχαριστώ. Taip, ačiū, gerimas pirmininkė. Taip noriu padėkoti pranešėjai už tikrai dokumentą reikia ναι, πάρα πολύ πλήρης εισηγήση του συντάκτη της έκθεσης και ελπίζουμε στο μέλλον θα έχουμε πολιτική αρτιότερη όσον αφορά τα δύο ευρωπαϊκά δίκτυα. Μέχρι σήμερα υπήρχε κατάτμιση, ε, δεν υπήρχε ευελιξία. Δεν πρέπει να φραφορτώνουμε τις ρυθμίσεις με λεπτομέρειες. Βέβαια θα πρέπει να υπάρχει εποπτεία από την Επιτροπή. Σωστά είναι αυτά που είπαμε για, τα, για τις ενεργειακές νησίδες. Και πάντα τα κριτήρια πρέπει να διέπονται από ευρωπαϊκό πνεύμα και εθνικό. Θα πρέπει βέβαια στην ε, ενεργειακή πολιτική που θα δημοφιλώσουμε στο μέλλον να ε, λάβουμε υπόψη τι ανανεώσιμε μορφέ ενέργεια και θα πρέπει η Κομισιόν να υπολογίσει το κόστο τη πυρηνική ενέργεια που σήμερα χρησιμοποιείται. Όχι μόνο την εκμετάλλευση και την κατασκευή, αλλά και το κόστος λειτουργίας. Γιατί ενδεχομένω τα ανανεώσιμα θα είναι κάτι το προτιμότερο.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 έγγραφο της Κομισιόν δεν έχει μια ευρεία προσέγγιση για τους ε, διαδρόμους ενέργειας και υγροποιημένου αερίου. Αυτό νομίζω θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε διάσκεψη κορυφή που μόλις έλεγε χώρα υπάρχει στα συμπεράσματα μια αναφορά Σύμφωνα με τα οποία θα πρέπει να υπάρχει διάκριση βάρος καμίας πηγής ενέργειας και εδώ έχω κατά νου κυρίως την διαφορά παραδοσιακών μορφών και μη παραδοσιακών. Α πούμε το αέριο ποσιστόλιθο θα πρέπει να τύχει της σωστής χρήσης γιατί θα πρέπει η Ευρώπη να εκμεταλλευτεί αυτή την πηγή αερίου στο μέλλον. 65 δισεκατομμύρια κυβικά εξορίγνονται στην Αμερική αυτό είναι πρέπει να το έχουμε υπόψη μας λοιπόν. Βέβαια η προοπτική αυτή είναι μακροπρόθεσμη αλλά αξίζει να μην την ξεχνάμε. Ευχαριστώ. Η κυρία Τικάου. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την έκθεσή του. Θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση για το μέλλον της ενεργικής πολιτικής της Ευρώπης θα έπρεπε να λαμβάνει υπόψη την εφαρμογή της ρήτρα της αλληλεγγύης που σχετίζεται με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Εάν ένα κράτος δηλαδή αντιμετωπίζει μια ενεργειακή κρίση, θα πρέπει οι άλλες χώρες μέλη να τον υποστηρίξουν. Η ενέργεια θα πρέπει επίσης να είναι προσβατή για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες το 30% του εισοδήματος μιας οικογένειας χρησιμοποιείται για την ενέργεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν η ενέργεια να παραμείνει προσιτή για τους πολίτες. Και όσον αφορά τώρα τη ρήτρα αλληλεγγύη, θα πρέπει να υπάρχουν αλληλοσυνδέσεις μεταξύ των κρατών μελών και να υπάρχουν ευφυή δίκτυα. Χρειαζόμαστε επένδυση της τάξης των 200 δισεκατομμυρίων ευρώ θα πρέπει λοιπόν να βρούμε τα απαραίτητα ε, χρηματοπιστωτικά μέσα για να το πετύχουμε. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να κοιτάξουμε κυρίως ε, πώς θα γίνουν πιο ε, ενεργειακά αποδοτικά τα κτίρια και επίσης να εξετάσουμε και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Για την ηλεκτρική ενέργεια θεωρώ ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τοπικά ανανεώσιμες πηγές που θα πρέπει να εντάσσονται σε ευφυή δίκτυα. Τελειώνοντας ε, έχω να πω ότι η Ήπεθρος αντιμετωπίζει ειδικά, ειδικές ανάγκες όσον αφορά την ενέργεια και θα πρέπει νομίζω να βασιστεί στις ε, ανανεώσιμες πηγές και θα πρέπει και δικά της δίκτυα να ενταχθούν στα ευρωπαϊκά ευφυή δίκτυα όταν εξετάσουμε τις νέες δημοσιονομικές προβλέψεις και το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα διαστατικά θαμεία, θα πρέπει να φροντίσουμε η ενεργειακή αποτελεσματικότητα να μην παραβλεφθεί και θα πρέπει να αποδώσουμε σημασία στις ανάγκες της ενεργειακής της υπαίθρου. Θα ήθελα να υποβάλω και μια ερώτηση στον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Υπάρχει μια δέσμη που προέβλεπε επενδύσεις για τα 10 επόμενα έτη. Θα ήθελα να ξέρω πού έχει προχωρήσει αυτό το πακέτο και αυτές οι επενδύσεις. Ευχαριστώ. στην Σχόλιο, ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πολύ <clears throat> τον εισηγητή για την παρουσίαση που μας έκανε και να σχολιάσω τρία σημεία. Καταρχήν, ο εισηγητή ανέφερε τις ευφυείς πόλεις και τη σημασία της ε, ε, ε, επάρκειας ενέργεια και η κυρία Τικάου επίσης το έθιξε αυτό μόλις με εντυπωσίασε, εγώ θεωρώ ότι είναι σημαντικό όταν μιλάμε για ανάγκε υποδομών να λαμβάνουμε υπόψη τις επιπτώσεις των μέτρων ενεργειακής επάρκειας όταν κρίνουμε ποιες θα είναι οι ανάγκες ολόκληρου των Ευρώπη και η, Ευρω... η μελέτη της ΕΚΟΦΗΝ για τις επιπτώσεις της εξοικονόμησης ενέργειας δείχνει ότι η εξοικονόμηση ενέργειας αντιστοιχεί σε 15 ναμπούκο. Πρέπει να το σκεφτούμε αυτό. Επίσης να σκεφτούμε την ιεραρχία και τα κριτήρια που ανέφεραν διάφοροι συνάδελφοι. Εγώ νομίζω πως εκτός από την προτεραιότητα του να εξασφαλίσουμε το να μην δημιουργηθούν ενεργειακές νησίδες, ε, να σκεφτούμε πολύ καλά τα κριτήρια και να σκεφτούμε επίσης και την αυξανόμενη σημασία του ηλεκτρισμού καθώς προχωρούμε και μήπως ε, ο εισηγητής θα μπορούσε αυτό να το λάβει υπόψη και το γεγονός δηλαδή ότι ο ηλεκτρισμός θα είναι προτεραιότητα ε, σε σχέση με άλλες μορφές ενέργειας. Και έπειτα για την αδειοδότηση είναι πρόσδεκτες οι προσπάθειες και η σημασία που δίνεται στην ανάγκη για εναρμόνιση. Θα πρέπει ωστόσο να εξασφαλίσουμε μια εναρμόνιση, ώστε το όριο αυτό να είναι το μάξιμο, ώστε στις χώρες όπου όντω προχωρήσει πιο γρήγορα η διαδικασία, να μην έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν να καταστήσουμε σαφέ ότι όσο πιο γρήγορα τόσο το καλύτερο και ότι η εναρμόνιση να είναι το μάξιμο όριο και όχι ένα μέσος όρος. Εκτιμώ λοιπόν πολύ τα όσα είπε ο εισηγητής. Ευχαριστώ. Γκίρεκ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ακούω την σημερινή συζήτηση. Και να σας πω που πραγματικά ότι λυπάμαι τον κύριο Βάγνερ. Γιατί είναι λες και ζητούσαμε από έναν ε, δικηγόρο να φτιάξει ένα αυτοκίνητο. Προσεγγίζουμε το θέμα δηλαδή από την πίσω πόρτα και η Ευρωπαϊκή Κομισιόν διευκολύνει τον εαυτό της βασικά. Δεν νομίζω πως ένας ε, δικηγόρος μπορεί να σχεδιάσει τα ευρωπαϊκά δίκτυα με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Εγώ νομίζω πως θα έπρεπε να είναι τελείως διαφορετική προσέγγιση. Να είμαστε δηλαδή πιο... Ε, αυστηροί και να συζητήσουμε για το ποια νομικά εμπόδια θα πρέπει να αποφύγουμε όσον αφορά τις νομοθεσίες συγκεκριμένων κρατών μελών. Σας εύχομαι λοιπόν κάθε επιτυχία στις προσπαθίες σας, παρόλα αυτά Πιστεύω πως δεν θα υπάρξει καλός προγραμματισμός και όπως με τις προηγούμενες προσπάθειες όλα αυτά θα καταλήξουν σε φιάσκο. Ταυτόχρονα συμφωνώ με την κυρία Μπομπίνσκα και με τον κύριο Κουάντρας ότι έχουμε αρκετή νομοθεσία. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι συγκεκριμένα προγράμματα. Ευχαριστώ. η και μετά άλλο ένα έχουμε Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι πάρα πολύ σύντομο. Καταρχήν, θα ήθελα να εκφραστώ όσον αφορά τη χρηματοδότηση. Θα πρέπει να διευκρινιστεί το θέμα αυτό και ε, έχω να πω ότι θα πρέπει ο συνάδελφο Σούζα Βάρκα να συμπεριλάβει και καινοτομικά σημεία όπω αυτά που ανέφερε η συνάδελφο Βαλεάν. Και θα πρέπει επίση να δούμε τι γίνεται με την ΕΙΜΠΕ που μπορούμε να έχουμε πολλαπλασιασμό, δεκαπλασιασμό θα έλεγα θα πρέπει να προσαρμόσουμε βέβαια τον προεπιλογισμό, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει σχέδια τα οποία ε, δεσμεύονται εδώ σε, ορισμένα, σε ένα ορισμένο πλαίσιο θα μπορούσαν να χρηματοδοτούν. Κατόπιν ε, συζητάμε για τη μεγάλη ιστορική αγορά, τους ε, διακανονιστές, αλλά η δυνατότητα αποθήκευσης μου λείπει εμένα, γιατί όλες οι θεωρίες του 2020 δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν εάν δεν έχουμε δυνατότητα αποθήκευσης του τις ενέργειες, ιδίω για τι ανανεώσιμες πηγέ ενέργεια και ίσω να δημιουργήσουμε και νησίδες. Ε, θα πρέπει να προχωρήσουμε προ αυτή την κατεύθυνση για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε αυτά τα καινοτομικά σημεία χρηματοδότηση. Πολύ σύντομα, συνάδελφο Καβάλιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συζητάμε μια έκθεση που είναι πολύ σημαντική για ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι πολύ σημαντικό ο συντονισμό με την έκθεση για τον μελλοντικό, τη μελλοντική χρηματοδότηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το μελλοντικό προπολογισμό. Όπω είπαν διάφοροι συνάδελφοι, Πρόκειται, χρειαζόμαστε, έχουμε ένα σύνολο μάλλον νομοθεσία ε, που είναι πλήρε και γι' αυτό το δώρο θα πρέπει να δούμε συγκεκριμένα προγράμματα, συγκεκριμένα για το ηλεκτρικό δίκτυο, ηλεκτρο, δίκτυο ηλεκτροδότησης και για το φυσικό αέριο που θα πρέπει να καλύπτουν ολόκληρη την Ευρώπη, να φροντίσουμε για την αποφυγή ενεργειακών νησίδων, αλλά να εξετάσουμε και το θέμα των νησιών, των ε, πραγματικών νησιών που έχουν πολύ ιδιαίτερα προβλήματα και θα πρέπει να μεριμνήσουμε για το θέμα των ευρωπαϊκών νησιών και των υποδομών για τα νησιά. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα να δώσω το λόγο στην Κομισιόν. Κύριε Μπενουά. Μάλιστα, σας ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ όλα τα μέλη της Επιτροπής σας για τις σημαντικές συμβολές τους σε αυτή τη τόσο σημαντική συζήτηση για την μελλοντική ενεργειακή υποδομή. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή γιατί πραγματικά στο έγγραφο εργασίας του θέτει όλα τα θέματα που διακυβεύονται αυτή τη στιγμή. Βέβαια γνωρίζουμε ότι χρειάζεται να δώσουμε σημασία σε όλους τους στόχους για το 2020 και ε, αποτελεσματική χρήση της ενέργειας και το θέμα των εσωτερικών αγορών συμμεριλαμβανούν και του Ευρωπαϊκού Συστήματος για την μεταβίβαση των, της ενέργειας της ηλεκτρικής ενέργειας καθώς επίσης και τους κανονισμούς για τους διακανονιστές. Υπάρχουν λοιπόν πολλά συγκεκριμένα στοιχεία για να ανάψουν μια πραγματική ευρωπαϊκή πολιτική υποδομή και αυτό νομίζω βρίσκει όλοι σας στην Επιτροπή σύμφωνη. Υπάρχουν τέσσερα θέματα πάρα πολύ σημαντικά για μας καταρχήν και το τονίσατε πάρα πολύ ωραία. Να έχουμε ένα κατάλογο καλών κριτηρίων για την επιλογή των σχεδίων και των προγραμμάτων. Εδώ θα είναι σημαντικότατος ο δικός σας ρόλος, ε, μια ιεράρχηση των κριτηρίων θα είναι οπωσδήποτε πάρα πολύ χρήσιμη για μας για να καταλήξουμε στην ε, εξέβριση των ε, προγραμμάτων που θα έχουν ευρωπαϊκό ενδιαφέρον. Κατόπιν είπατε ότι θα πρέπει να επιταχυνθεί η διαδικασία διαδότησης. Δεν παραβλέπουμε τη στάση του πληθυσμού, το έχουμε κατά νου ε, και αυτό συνδέεται συγγνώμη, και με τη χρηματοδότηση γιατί όσο πιο πολύ καθυστερούμε τόσο πιο ακριβή θα είναι η διασύνδεση. Πρέπει λοιπόν να βρούμε από κοινού λύσεις για την έγκριση, για τη χρηματοδότηση και για τη χρηματοδότηση θα βασιζόμαστε στις αγοράς. Αυτή είναι η προσέγγιση και όπως ελέγχθη από διάφορα μέλη κατά πάση όταν δεν θα είναι αρκετό όταν θα πρέπει να εξετάσουμε την ασφάλεια της τροφοδότησης και αναφερθούμε στην πλήρη ε, ολοκληρώση των αγορών. Πάνω σε αυτά λοιπόν θα χαιρετίζαμε τις όποιες συμβολές σας που πάντα είναι πολύ χρήσιμες. Δύο τελευταία χρόνια σημειώνουμε το θέμα των προτύπων. Είναι κάτι όμως που συζητήθηκε στο χρονοδιάγραμμα του 2050 και δεν σχετίζεται με τη συζήτηση τη σημερινή και όσον αφορά τους ε, τόπιους, ε, ε, τις τόπιες πηγές άκουσα ότι ελέγχθη για το μη παραδοσιακό φυσικό αέριο. Δεν χρειάζεται νομίζω να τσακωθούμε και εδώ γιατί αυτό είναι για το 2080. Αλλά οπωσδήποτε καλό είναι να εξετάσουμε το θέμα των ε, εκάστοτε τοπικών ε, αποθεμάτων. Γιατί θα πρέπει να καταλαβαίνουμε αυτό που έχουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σα ευχαριστώ για τη συμβολία σα και περιμένουμε να ακούσουμε τι μελλοντικέ συζητήσει του θέματο εδώ. Ε, και εγώ σας ευχαριστώ. Λόγω του προχωρημένου της ώρας ε, θα κλείσουμε εδώ τη συζήτηση. Το επόμενο σημείο θα το εξετάσουμε μετά τη Ζεφορία, Αν συμφωνείτε θα προσπαθήσουμε να ψηφίσουμε στα γλίγορα για να μπορούμε να περάσουμε και γλίγορα και στην ακρόαση. Έχετε όλες τις κάρτες σας. Όχι, ναι nice research. Ja, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, μ' ακούτε, με καταλαβαίνετε. Ε, Unterhaltungsprogramm. Ή έχουμε τα παιδιά παίζει τώρα. It's possible that we can... Λοιπόν, äh, äh, Τροπή του κανονισμού του 462.000 ε, Ευρωπαϊκού Κοινωνικού του Συμβουλίου για τη Δημιουργία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων Πληροφοριών ω προ τη διάρκεια του. Μία ψηφοφορία. Τελική ψηφοφορία αμέσω. Ποιο είναι υπέρ. Ηλεκτρονικά μάλλον. Λοιπόν, ηλεκτρονικά, με συγχωρείτε, επειδή είναι τελική ψηφοφορία, πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά. Doesn't work, huh? Wonderful, it doesn't work. Α, δεν λειτουργεί το σύστημα, πολύ ωραία. Alessandra. Try. The vote is open. ψηφοφορία. Λειτουργεί ή δεν λειτουργεί. Ε, όχι με ανάθεση του τότε. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ με ανάθεση χειρός. Κλαπς. 41 für. 41 dafür. 41 υπέρ. And plus Miss Merkel, okay. Alles einstimmig so beschlossen. Λοιπόν, αποφασίστε αυτό ομόφωνα. Επόμενο σημείο. Έκθεση Μπέλετ. Ποιο είναι τη συμβαστική 1. Με ανάθεση χειρό παρακαλώ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Συμβαστική 7. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 46 καταπίπτει. Συμβαστική 8. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 18 καταπίπτει 9 συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 με προφορική τροπολογία ποιος είναι υπέρ κατά αποχές ευχαριστώ εγκρίνεται Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 16 με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ Ξέχασα κάτι. 21 καταπίπτει. Κατέπεσε. Λοιπόν, συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 44. Σε δύο τμήματα. Με προφορική τροπολογία στο πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 κατά 29 35 32 συγγνώμη 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 37 muss gemacht werden? Ah, την 37 πρέπει να ψηφίσουμε. Ε, ναι. Λοιπόν, 37. 37 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 42 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ένα λεπτό. Τι τρέχει. Εντάξει, εντάξει είμαστε. Τελική ψηφοφορία. Άρχιτη ψηφοφορία. Α, ηλεκτρονικά είπαμε δεν γίνεται. Γίνεται. πέρασε ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια σε όλου του συζητητέ και εκείνου που εργάστηκαν τόσο πολύ για αυτά τα θέματα. Περνάμε τελειώσαμε τι ψηφοφορίε. zum nächsten Punkt, nämlich zum Tagesordnungspunkt Derivatezentrale. Περνάμε τώρα στα παράγωγα κεντρικούς αντισυμβαλόμενους και κεντρικά μητρών συναλλαγών. We have done. No, we did two No, we have done the village. We have done. Huh? Yeah. Was, was...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 Uh, uh, Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, συνάδελφοι. Μου το σχέδιο κανονισμού για την εποπτεία των παραγόγων είναι μια υποχρέωση που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην συνεδρίαση των G20 όταν αποφασίστηκε να επεκταθεί ο κανονισμός στις, δημοσιονομικές χρηματοπιστωτικέ αγορές ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και ρύθμιση των αγορών αυτών. Ο κανονισμός αυτός ήδη επηρεάζει τη ΣΥΠΑ ω αποτέλεσμα αυτή τη συμφωνία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Κομισιόν επέκτηνε έκανε μάλλον ε, μακρές διαβουλεύσεις και το σχέδιο που έχουμε είναι το αποτέλεσμα όλης αυτής της προεργασία που έγινε πριν έρθει το σχέδιο κανονισμού στο Κοινοβούλιο. Τώρα, γιατί συμμετέχει η Επιτροπή μας και γιατί ζητήθηκε η γνωμοδότηση από εμά στη συζήτηση. Όταν μιλάμε για τα παράγωγα και, και παρόμοια είδη χρηματοπιστωτικών μέσων δεν χρησιμοποιούνται μόνο από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αλλά και από μη χρηματοπιστωτικές εταιρείες επιχειρήσεις και γι' αυτό και εμεί ζητήσαμε να γνωμοδοτήσουμε. Υπάρχουν διάφορα θέματα λοιπόν που σχετίζονται με επιχειρήσεις που, ε- που λειτουργούν στον τομέα το εμπορίο αγαθών, τροφίμων, ε, δημητριακών, ε, μετάλλου, ηλεκτρισμού και χρησιμοποιούν αυτά τα παράγωγα για να προωθήσουν τις επιχειρήσεις τους. Επίση, αυτά τα μέσα χρησιμοποιούνται ευρύτατα από διάφορα είδη επιχειρήσεων, κυρίως τις μεγάλες εταιρείε, για να μειώσουν τους ε, οικονομικούς κινδύνους ή εν πάση περιπτώσει να αναχαιτήσουν κινδύνους που αντιμετωπίζουν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους. Επειδή χρησιμοποιούνται λοιπόν για την ε, διαχείριση ή επειδή χρησιμοποιούνται για την αγορά των αγαθών, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μέσα τα οποία είναι απλά και μόνο κερδοσκοπικά και ότι χρησιμοποιούνται από τις εταιρείες ε, πολύ συχνά αποσπασμένα από τα υπόλοιπα στοιχεία κυριότητας των εταιριών. Αυτά τα παράγωγα λοιπόν ε, όταν χρησιμοποιούνται έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο από τις εταιρείες αυτές δεν δημιουργούν συστημικό κίνδυνο. Αυτό είναι μεγάλο ε, ανησυχία των ρυθμιστών και γι' αυτό και θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας πιστεύω στην αντικειμενικότητα των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων και τους, και τους καταναλωτές. Πολύ ενδιαφέρουσα ακρόαση δεν είχαμε με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας ενέργειας και των οργανώσεων των καταναλωτών όπου εκφράστη μια πολύ έντονη άποψη σε σχέση με αυτό το σχέδιο κανονισμού. Εν γέννη πιστεύω πως το σχέδιο κανονισμού ε, δίνει περισσότερο η διαφάνεια και λιγότερο κίνδυνο, αλλά όταν μιλάμε για το συγκεκριμένο είδος εταιριών, δηλαδή μη ε, χρηματοπιστωτικά εταιρείε, πρέπει να βρεθεί η σωστή ισορροπία ανάμεσα στην υπερβολική ρύθμιση, τη σωστή ρύθμιση και την δυνατότητα αυτών των εταιριών να έχουν πρόσβαση στα χρηματοπιστωτικά μέσα που μειώνουν τον κίνδυνο που διατρέχουν στις κανονικές τους δραστηριότητες. Εξετάζοντας λοιπόν και βλέποντας από την άποψη της δικής μας Επιτροπής το σχέδιο κανονισμού, ακριβώς αυτό είναι το θέμα. Πού πρέπει να τεθεί η ισορροπία ώστε να υπάρχει με μεγαλύτερη διαφάνεια, αλλά ταυτόχρονα να δίνεται ευκαιρία στις εταιρείε, κυρίως στις μικρότερες, να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα χρηματοπιστωτικά μέσα. Εγώ πρότεινα διάφορα πράγματα εδώ Ταυτόχρονα να σας πω ότι η προθεσμία για τη συζήτηση έχει παραταθεί, ώστε θα έχουμε λίγο παραπάνω χρόνο για να εξετάσουμε πιο προσεκτικά το έγγραφο πριν να υποβάλουμε την πρότασή μας και τη γνωμοδότησή μας στην αρμόδια της Επιτροπής που είναι η ΕΚΟΝ. Να σας αναφέρω επίσης τροπολογίες που εγώ θα πρότεινα να λάβετε υπόψη σχετίζονται με την αποσαφήνιση της διαδικασίας την διευκρίνηση κάποιων ορισμών, την διαφανέστερη εποπτεία και πιο προβλέψιμη εποπτεία βια τις εταιρείες, να αποφευχθεί το σοκ ε, συμψηφισμού, όπου σημαίνει ε, τις μικρές εταιρείες που πηγαίνουν σε κάποιο οίκο συμψηφισμού, που σημαίνει χρόνο και χρήμα. Θα πρέπει αυτό δηλαδή να μπορεί να βληθεί ώστε να μην να αποφευθεί το σοκ για τους μικρούς χρήστες αυτών των μέσων. Και έπειτα έχω και κάποιες τροπολογίες που θέλω να λάβετε υπόψη σας, να μελετήσετε και αφορούν κάποιο είδος διαπλοποίησης στη διαδικασία, ιδιαίτερα για εταιρείε που δεν είναι χρηματοπιστωτικές και όπου η υπερβολική ε, ρύθμιση σημαίνει πολλές περισσότερες δαπάνες που τελικά αντικατοπτρίζονται στις τελικές τιμές στον καταναλωτή. Αυτό είναι το ζουμί των τροπολογιών που σας προτείνω. Προσβλέπω στη συζήτηση μαζί σας και στις δικές σας, στη δική σας συμβολή και να σας πω και πάλι φαίνεται ένα πολύ τεχνικό θέμα να είναι, αλλά επηρεάζει τις ε, τιμές του καταναλωτή για πολύ, πολλά αγαθά. Και από την άλλη πλευρά επηρεάζει και τις δυνατότητες των καταναλωτών να παρακολουθούν διαφανώς τι συμβαίνει στην αγορά, να επηρεάζουν τον ανταγωνισμό και τις τιμές. Έτσι, επίσης, δίνεται μεγαλύτερη δυνατότητα στον, στον ρυθμιστή, ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Αρχή Εποπτείας των Αγορών, να παρέμβει και να ε, εκτιμήσει ευρύτερα τους κινδύνους ε, που διέπουν την αγορά, κάτι το οποίο πιστεύω πρέπει να υποστηρίξουμε πλήρως. Σας ευχαριστώ πάρα κύριε Καλφίνη για τόσο ακριβή αυτή η εισαγωγή. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στους συναδέλφους. Πρώτος είναι ο κύριος Μπένσιν. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστώ τον κύριο Κάλφιν για την τόσο καλή εργασία του. Γενικά Χαιρετίζω την προτινόμενη νομοθεσία από την Κομισιόν, γιατί προφανώ χρειάζεται διακανονισμό για εκείνα τα χρηματοπιστωτικά ε, Ινστιτούτα που οδήγησαν στην οικονομική κρίση. Βέβαια είναι γνωστό ότι δεν μπορούμε τα ίδια φάρμακα να χρησιμοποιήσουμε για όλους γιατί κάθε κράτος έχει διαφορετικό προφίλ κινδύνου. Η περισσότερες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τα παράγωγα για να καλύψουν κινδύνους που υπάρχουν από τις άλλες τους ε, συναλλαγές. Απορρισματική διαχείριση του κινδύνου σημαίνει ότι προσπαθούν να καλύψουν με τα παράγωγα και ο, ο κανονισμός αυτός θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στις αγορές ενέργειας και θα παρεμποδίσει την εξέλιξη επαρκών και αποτελεσματικών αγορών ενέργειας στην Ευρώπη. Και γι' αυτό χαίρομαι που η Επιτροπή μας αποφάσισε να γνωμοδοτήσει το θέμα αυτό για να είμαστε σίγουροι ότι οι αγορές ενέργειας δεν θα υποφέρουν από υπερβολικές διατάξεις. Δεν νομίζω ότι οι αγορές ενέργειας οδηγούν σε ένα συστημικό κίνδυνο. για το, να διακανονίσουμε ε, τον κανονισμό για την νομοθεσία μάλλον για τα OTC χωρίς να λάβουμε υπόψη μας τις πτυχές ε, που σας προανέφερα δεν θα έχουμε το σωστό αποτέλεσμα. Χαίρομαι που λαμβάνετε υπόψη σας ε, τις ειδικές προϋποθέσεις που διέπουνε της ε, εταιρείας ε, παραγωγής και προμήθειας ενέργειας. <coughs> Θεωρώ ότι υπάρχουν ορισμένα σημαντικά θέματα που θα πρέπει να μην παρευλέψουμε στην έκθεση του μας. Παραδείγματος χάρη το εμπόριο μεταξύ των ομάδων θα πρέπει δηλαδή να είναι δυνατόν να υπάρχει μια εξαίρεση στην περίπτωση που οι συναλλαγές γίνονται με θηγατρικές εταιρείες. Πολλές φορές προσπαθούν με, ένα παράγοντα οι επιχειρήσεις αυτές σε ένα όμιλο να αποφύγουν ένα μεγαλύτερο κίνδυνο. Επίσης, οι εξαιρέσεις για τις συναλλαγές μεταξύ των μελών μιας ίδιας ομάδας λαμβάνονται υπόψη σε άλλους τομείς, όπως το Μάιφλ, παραδείγματος χάρη. Επίσης υπάρχει ανάγκη διακανονισμού για τις εταιρείε ενέργειας. Εάν δεν ξεπερνάμε ένα κατόφλι clearing, δεν θα πρέπει να περνάνε απαραίτητο σε clearing των ε, παραγόγων τους, επειδή ο εταίρος τους είναι, ανάλογα δηλαδή κατά πόσο εταίρος τους είναι χρηματοπιστωτικό Ιστιτούτο ή όχι. Θα πρέπει να υπάρχουν κατόφλια, αλλιώς θα υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις με ενεργειακέ επιχειρήσεις οι οποίε θα έχουν πολλές συναλλαγέ με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Περιτά. Ευχαριστώ. Η συνάδελφος βαλιαν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον εισηγητή. Γιατί εισήγηση που μας έκανε. Περιμένουμε ένα έγγραφο στο οποίο να εργαστούμε. οι κίνδυνοι που συνδέονται με την έκρηξη των χρηματοπιστωτικών αγορών και των παραγωγών είναι, αποδεικνύουν ότι πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά και αυτό είναι μια απαραίτητη ε, προϋπόθεση. Αυτό που πιστεύω είναι ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε ισορροπημένη προσέγγιση. Καμία οικονομία δεν μπορεί να ανθίσει αν κανείς δεν θέλει να αναλάβει τον κίνδυνο η χρηματοδότηση ενός προγράμματος εξαρτάται από το αν κάποιος είναι έτοιμος να φέρει τον συνδεόμενο κίνδυνο και είναι καλύτερο να μοιράζονται οι κίνδυνοι. Τα παράγωγα είναι καλά για την μοιρασιά ή την ανακατανομή του κινδύνου και γι' αυτό και τα παράγωγα θα πρέπει να μπορούν να είναι κομμένα και ραμμένα στις ανάγκες των χρηστών. Ωστόσο, ε, οι αυξημένε συναλλαγές σε OTC θα πρέπει να, ακολουθείτε και, ε, θα να ακολουθούνται από μεγαλύτερη διαφάνεια γιατί είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε το κίνδυνο της ε, αδυναμίας κάλυψης από τον εταίρο. Δεν είναι εύκολο πάντοτε να, δει κανεί την πιθανότητα αδυναμίας αποπληρωμής ενός χρέους. Είναι δύσκολο να δούμε πώς δημιουργείται ένα δίκτυο μηβαίας εξάρτησης που είναι πολύ δύσκολο κανείς να το ε, αποδομήσει και να το αντιληφθεί πώς λειτουργεί. οι ρυθμιστές μέχρι σήμερα δεν μπόρεσαν να εντοπίσουν τους κινδύνους ε, ε, Γι' αυτό και υπήρξαν τόσο σημαντικές συνέπειες για την ε, χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Ε, συμφωνώ λοιπόν ότι τα βασικά στοιχεία που προτείνει η Κομισιόν, καταρχήν ένα κεντρικό μητρό για τη συλλογή των στοιχείων, ιδιαίτερα για τους όγκους και τις τιμές, με στόχο την αύξηση της διαφάνειας και την επιχειρηματική, ε, τη λειτουργική μάλλον αποτελεσματικότητα της αγοράς και δεύτερον έναν ε, γραφείο συμψηφισμού για τους κεντρικούς αντισυμβαλόμενους. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να, τα διαχειρι... να, να γίνεται πολύ επαγγελματική διαχείριση και επίσης τα όσα είπα για τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα που υπάρχουν μάλλον για την ε, βιομηχανία ενέργειας, όπου πιστεύω θα πρέπει να γίνει διάκριση όχι μόνο για την ενέργεια, αλλά και για διάφορους άλλους οικονομικούς τομείς, γιατί φυσικά είναι προφανές ότι η αποτυχία μιας εταιρείας δεν θα οδηγήσει εκεί σε κατάρρευση της αγοράς και στο εφέ ντόμινο. οι συμβάσεις των παραγόγων μπορεί κάποιες φορές να οδηγήσουν σε επιφόρτιση της αγοράς χωρίς λόγο, ενώ με μεγαλύτερη διαφάνεια μπορεί να υπάρχουν ειδικά προγράμματα, μάλλον προϊόντα OTC, τα οποία θα είναι όμως υποέλεγχο και τα οποία θα είναι συγκεκριμένα για τη διαχείριση της κάθε εταιρείας. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να ρυθμιστούν βέβαια οι χρηματοπιστωτικές αγορές, ενώ θα διατηρηθεί η ευελιξία, η δυνατότητα για την καινοτομία και επιλογή. Äh, Σας ευχαριστώ πολύ. Κανένας άλλος δεν έχει δει στον Δεν ξέρω, ο κύριος Κάλβιν θέλει πάλι το λόγο. Όχι. Ναι, Παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ. Ήθελα να πω μία πρόταση. Θα ήθελα να ευχαριστώ τους συναδέλφους που τοποθετήθηκαν πάνω στο θέμα αυτό. Πραγματικό πιστεύω ότι κινούμεθα προς την ίδια κατεύθυνση και είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε πολύ καλή γνωμοδότηση τελικά από την Επιτροπή μας. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στις 2 Μαρτίου έχουμε την υποβολή για τις τροπολογίες. Λοιπόν, κλείνουμε αυτό το σημείο της μερικής διάταξης ευχαριστώντας όλους τους συναδέλφους και αμέσως θα προχωρήσουμε μετά από ένα σύνομο διάλειμμα με την ακρόασή μας. Δύο λεπτά διάλειμμα. König. Doch. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, noch einmal alle ganz herzlich begrüßen. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους στην μήνυ ακρόαση. Ξέρετε ότι το θέμα της καινοτομίας είναι πάρα πολύ σημαντικά για μας όσον αφορά τη δυνατότητα βιβλίου στο μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συνάδελφος Μέρκης είναι εδώ στα αριστερά μου Τυχαίο βέβαια αυτό. Να το κάθε αριστερά. Είναι υπεύθυνη συγγήτρια για το τομέα. Και μας είχε προτείνει να ακούσουμε κάποιους υπερογνώμονες. Δεν θα να ευχαριστήσω όλους τους υπερογνώμονες που είναι εδώ. Και μία μικρή παράκληση. Εγώ δεν θα μιλήσω πέντε λεπτά, δύο θα μιλήσω. Αν όλοι αντί να μιλήσετε 15 λεπτά, μιλήσετε 10, θα έχουμε περισσότερη δυνατότητα οι συνάδελφοι να υποβάλουν ερωτήσεις, πράγμα που θα ήταν χρήσιμο για όλους. Λοιπόν, ίσως όλοι μπορείτε να είσαστε πιο σύντομοι. Αν ο καθένας μπορεί να μιλήσει 10 λεπτά, θαυμάσια. Αυτά. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Μέρκες για να κάνει κάποια εισαγωγή, αν θέλει. Thank you, Chair. Uh, actually, going to follow your Εγώ θα ακολουθήσω το παράδειγμά σας, το λαμπρό, και θα είμαι σύντομη, πάρα πολύ σύντομη. Ενδιαφερόμαστε όλοι πάρα πολύ για το θέμα της καινοτομίας. Και μας ενδιαφέρει να δούμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε την καινοτομία ως μια κινητήριο δύναμη στην Ευρώπη για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και ταυτόχρονα να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί. Πραγματικά ανυπομονώ να ακούσω τις παρεμβάσεις και τις ερωτήσεις των συναδέλφων ώστε να έχουμε μια ζωντανή συζήτηση για το πώς θα λειτουργήσει η, η καινοτομία <laughs> πώς θα είμαστε συγκεκριμένοι και πώς η στοχοθεσία μπορεί να καθοδηγήσει και να δώσει όθηση και στην καινοτομία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα καταρχήν να δώσω το λόγο στον δόκτωρα Πέτερ Κότερ, ε, διευθυντή QTI Innovation Europe, Arco Consult. Κανένα άλλο δεν θέλει το λόγο. Ωραία. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Good morning. Καλημέρα σας. Λέω κύριος Κόταλ. Είναι μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι εδώ, διότι έχω την ευκαιρία μαζί σας να μοιραστώ αυτή μου την ταπεινή άποψη όσον αφορά την καινοτομία σε σχέση με τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ονομάζομαι Πέτερ Κόταλ και ε, τώρα είμαι μάνατζερ σε δύο τέτοιες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και έχω διατελέσει ερευνητής αλλά και εκτελεστικό στέλεχος σε μεγάλες εταιρείε, αλλά είμαι και επιχειρηματίας. Πάρα πολύ με ενδιαφέρει η καινοτομία και αν μου επιτρέπετε έχω να σας εκθέσω κάποιες απόψεις. Πρώτα πρώτα δύο λόγια για το τι κάνουμε. Όπως σας είπα τώρα έχω δύο μικρομεσαίες επιχειρήσεις και έχουμε επικεντρώσει τον ενδιαφέρον μας στην, ε, σε, σε πρωτοπόρες ε, τεχνολογίες και προσπαθούμε να δούμε πώς με καινοτόμες επιχειρήσεις θα προχωρήσουμε ούτω ώστε να τα καταφέρουμε καλύτερα στην ε, αγορά. Στην παγκόσμια αγορά και πριν από λίγα χρόνια είχαμε τον πρώην Ουκρανό πρόεδρο που με διοξίνη είχε, α, υποστεί κάποια επίθεση και ήταν και αυτός σε εκείνη την επιχείρηση ε, ασθενής μας. Και επομένως μας ενδιαφέρουν οι νέες τεχνολογίες για να δούμε επίσης πώς θα μπορούμε να αναπτύξουμε και κάποιες στρατηγικές καινοτόμες απλή στρατηγική προσπαθούμε να ελκύσουμε συνεταίρους στον ιδιωτικό τομέα και να έχουμε ένα κέντρο καινοτομία κάτι το οποίο ανάγεται στην ε, πλατφόρμα που θέλουμε να φτιάξουμε Και έτσι προσπαθούμε να επιφέρουμε κάποιες ε, μεταρρυθμίσεις επιτυχής. Ο βέβαια το κρίσιμο θέμα εδώ είναι η χρηματοδότηση. Γιατί πολλοί θα μπορούσαν να πούνε ότι ε, το πρόγραμμά σας δεν αξίζει χρηματοδότηση. Όμως έχουμε και εναλλακτικά προγράμματα. Και γι' αυτό από δική μας πλευράς θεωρούμε ότι άπαξ και κανείς χαρακτηρίζει ένα πρόγραμμα καινοτόμο, ότι αφορά την καινοτομία, τότε διατρέχει κίνδυνο να μην ελκύσει χρηματοδότηση. Τι είναι μικρομεσαία επιχείρηση. Οι ιδέες να γίνονται προϊόντα και υπηρεσίες. Και επίσης η μία τέτοια επιχείρηση ενώνει, γεφυρώνει πάρα από το κενό που υπάρχει μεταξύ πανεπιστημίων και βιομηχανίας. Βεβαίως το κίνητρο εδώ είναι σημαντικά κέρδη. Τώρα βέβαια υπάρχουν και μεγάλες επιχειρήσεις στην υπόθεση της καινοτομίας, υπάρχει κρατική έρευνα. Αυτή όμως δεν διατρέχουν κανένα ρίσκο, αντίθετα με τις ΜΜΕ. Επομένως, μπορείτε να δείτε τώρα τα, ποια αυτά είναι, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ρόλου της ΜΜΕ για την καινοτομία. Επίσης, έχουμε μια άλλη συμβολή των ΜΜΕ, το ότι πρέπει να επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στο εμπόριο, στο επιχειρήν. Χρειάζεται πνεύμα συνεργασίας γιατί εξαρτώνται και από άλλους και από τους άλλους εμπλεκόμενους στην αλυσίδα της διαδρομής της καινοτομία. Για να δούμε τώρα τι γίνεται με τις ευκαιρίες που προκύπτουν και τι γίνεται και με τους άλλους που ασχολούνται με την καινοτομία. Είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει χρηματοδότηση για έρευνα και ανάπτυξη. Αλλιώς δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει κανείς αυτή τη διαδρομή για να ζήσει καινοτομία. Να μην σταθούμε περισσότερο σε αυτό. Γιατί αυτό θα το καλύψει κάποιος άλλος από τους προσκεκλημένους ομιλητές. Κάτι άλλο τώρα είναι το κατά πόσον έχουμε πρωτοπόρες ε, επιχειρήσεις που να εκμεταλλεύονται τις ιδέες από τα πανεπιστήμια. Και έτσι να γίνονται πιο ανταγωνιστικές. Ε, τελικά είναι πάρα πολύ σημαντικό, περισσότερο από όλα σημαντικό αυτό το να υπάρχουν τέτοιε πρωτοπόρε τάσει και ιδέε. Ανθρώπινη πόρη τώρα. Αν δει κανεί τι γίνεται στην αγορά, είναι πάρα πολύ δύσκολο κανεί να βρει κάποιον που να έχει τι κατάλληλε δεξιότητε, ούτω ώστε να δουλέψει στον τομέα τη καινοτομία και να πει ότι κάποιο είναι <clears throat> ερευνητή αλλά και επιχειρηματία. Αυτό ίσω είναι θέμα του εκπαιδευτικού συστήματος. Αν κάνει θέλει να προχωρήσει προς την ε, καινοτομία, χρειάζεται να φτιάξουμε μια καινούργια γενιά από ερευνητές και επιχειρηματίες. Ταυτόχρονα. Ε, φυσικά και χρειάζεται συνεργασία ιδιωτικού και δημοσίου τομέα γιατί όταν πάβει χρηματοδότηση τότε πολλές φορές πάβει και η διαδρομή αυτής της επιχείρησης αλλά ε, θα πρέπει να το δούμε αυτό το πρόβλημα γιατί ισχύει αυτή η συνεργασία μόνο πρόθεσμα. Τώρα όσον αφορά το μη ενιαίο του περιβάλλοντος στο επιχειρήν ή το, το πολύπλοκο ε, περιβάλλον. Το υπερβολικά πολύπλοκο κάτι το οποίο είναι αποθαρρυντικό, είναι κάτι το οποίο υπονομεύει, δυναμητίζει τις ΜΜΕ. Δεν είναι δυνατόν να ευνοείται η διαδρομή μιας επιχείρησης όταν το περιβάλλον είναι υπερβολικά περίπλοκο. Άρα και εδώ θα πρέπει να προβληματιστούμε. Ας πούμε ε, ένα παράδειγμα από τη βιομηχανία μπορεί να είναι οι μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες όποτε βλέπουν την ευκαιρία τότε κάνουν τη δική τους διαδικασία παραγωγής. Αυτό όμως δεν μπορεί να το κάνει ΜΜΕ ε και το ίδιο ισχύει βέβαια και με την περιπλοκότητα της νομοθεσίας. Τώρα, όλοι οι μπλεκόμενοι στην καινοτομία θα πρέπει να συνεργάζονται, θα πρέπει να υπάρχει κάποιο είδου συνένεση. Να υπάρχει επίσης ένα επιχειρηματικό πνεύμα. Αυτό χρειάζεται οπωσδήποτε. Θα πρέπει κανείς επίσης να έχει εκπαιδευτεί ούτως ή να αποδέχεται την αποτυχία, κάτι το οποίο συμβαίνει πολλές φορές στην προσπάθεια για καινοτομία. Επομένως θα πρέπει, ανεξάρτητα από το αν λέμε κάτι καινοτόμο ή όχι, μια προσπάθεια, θα πρέπει να επικεντρώνουμε την προσοχή μας στο αποτέλεσμα. Θα πρέπει επομένως το περιβάλλον να βοηθάει την ε, προσπάθεια καινοτομία, θα πρέπει να έχουμε ε, πρωτοπόρες προσπάθειες για καινοτομία που να είναι και ανταγωνιστικές. Επίσης θα χρειαζόμαστε μέτρα και πιλωτικά προγράμματα ούτω ώστε το, το, το, όλο δίκτυο καινοτομία στην Ένωση να ανανιώνεται, να ξανανιώνει. Ε, επίσης θα πρέπει κανείς να θεωρεί την καινοτομία κάτι σαν τέχνη. Δεν είναι δουλειά, είναι αποστολή. Δεν είναι κανείς να αναγκάσει κάποιον να προσπαθήσει να είναι καινοτόμος, Ούτε είναι το να, να υποστεί ε, ρύθμιση υπερβολική. Ε, θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχο λοιπόν περιβάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση και χρειάζεται ε, μια ομάδα αρμονική που να έχει κατάλληλη ηγεσία. Ευχαριστώ. Δόκτωρα Κόταλ, δέσω το λόγο στον δόκτωρα Άχατσα, που είναι αντιπρόεδρος της Siemens και επικεφαλής της έρευνας και ανάπτυξης στη Siemens. Sehr geehrter Herr Reul, vielen Dank für die Einladung. Thank you very Κύριε Ρόλη, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή Σα Ευχαριστώ που μου δίνετε δυνατότητα να σα μιλήσω εδώ. Αυτό που θα ήθελα να κάνω θα ήταν να ορίσω στα γλίγορα το ότι είναι η κοινωνία πρωτού αρχίσω την παρουσίασή μου. Ο ορισμό μου είναι παρόμοια με τον ορισμό του Πίτερ Κότολ. Δηλαδή λέμε έχει δύο πτυχέ. Η μία πτυχή είναι η ιδέα, η άλλη πτυχή είναι οι ιδέες αυτές να περάσουν στην αγορά. Και αν η ιδέα δεν ήταν επιτυχή στην αγορά, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Δηλαδή, καινοτομία είναι η ιδέα εφαρμογή στην αγορά. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική η καινοτομία για εταιρείε όπως τη Siemens. Και άμα να δούμε ποια είναι η διαφοροποίηση για μια επιχείρηση να είναι πιο φτηνή, έχει την καλύτερη οργάνωση πώληση. Η ΣΥΜΕΣ είπε ότι εμεί θέλουμε να είμαστε οι καινοτόμοι. Να είμαστε δηλαδή πρώτοι στην αύξηση της ανταγωνιστικότητα στην δημοσιογεία και σε ευφυείς λύσεις. Αυτό είναι κάτι καινούργιο για μια εταιρεία όπως η Siemens γιατί πριν από στα 160 χρόνια που υπάρχει η, η είχε έχει αλλάξει την προσέγγιση της και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Εφορία για πολλούς σημαίνει ότι είμαστε φιλικοί προς το περιβάλλον, αλλά νομίζω ότι άμα θέλει να είναι κανένα 160 χρόνια και πάνω σε επιχείρηση, δεν θα πρέπει αρκεί μόνο να είναι φιλική προς το περιβάλλον. Θα πρέπει επίσης να είναι αηφόρο όσον αφορά το προσωπικό, α πούμε, όταν αφορά του ανθρώπου. Όταν συζητάμε τι δραστηριότητε μα έρευνα, θα πρέπει να δούμε ποιε είναι οι προκλήσει που πρέπει να επιληθούν. Και γι' αυτό αναφέρομαι εγώ στι μεγάλε προκλήσει, όπω έχουμε ορίσει, και θα επανέλθω σε αυτό το θέμα. Περισσότεροι εγκαταλείπων, εγκα, φύστανται συγγνώμη στις πόλεις. Το 2007 ήταν η πρώτη χρονιά που περισσότεροι ζούσαν στα αστικά κέντρα από ότι στην Ήπεθρο. Οργάνωση λοιπόν είναι ένα σημαντικό σημείο, αλλά και το θέμα των προκλήσεων για τις υποδομές, οι μεταφορές, ε, οργάνωση λοιπόν γενικά είναι ένα δεδομένο. Μια άλλη πρόκληση, μια άλλη τάση αν θέλετε, είναι οι δημογραφικές αλλαγές. Ε, δηλαδή υπάρχει γύρινση του πληθυσμού, καλό για το κάθε άτομο, αλλά αυτό αλλάζει και τροποποιεί την κοινωνία. Και όσον αφορά την προστασία της υγείας, το περιβάλλον θα πρέπει να προσαρμοστεί στους ε, ηλικιωμένους. Και αυτό λοιπόν είναι μια αλλαγή που πρέπει να έχουμε κατά νου. Κατόπιν, κάποια εποχή συζητεί το κατά πόσον υπάρχει κλιματική αλλαγή ή όχι. Τώρα δεν υπάρχει πια αμφιβολία και συζήτηση. Υπάρχει. Αλλά θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και αυτή μια μεγάλη πρόκληση λοιπόν. Και η τέταρτη που έχουμε κατά νου είναι η παγκοσμιοποίηση. Όταν μπορούσαμε να εργαστούμε και να δρούμε ε, τοπικά, στο παρελθόν η κατάσταση διαφορετική. Τώρα δεν ισχύει αυτό όμως πια. Τώρα κινούμεθα παγκόσμια και οι επιχειρήσεις και η έρευνα. Πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε με τους ε, οι ε, γειτονέ μα στην, ε, στην ε, Ασία, στην, Αμερικανού. Λοιπόν, δεν είναι πια ο παλιό κόσμο που ξέραμε, είναι καινούριο κόσμο που έχει αλλάξει ριζικά. Και εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι κανένα ανοιχτό. Ακολουθούμε δηλαδή την ιδέα τη ανοιχτή καινοτομία. Εξακολουθούμε να έχουμε δηλαδή τις ερευνητικέ μας δραστηριότητε στις Ζήμε. Έχουμε πάνω από 2.000 ερευνητέ και στην Ευρώπη και ανά τον κόσμο αλλά ξέρουμε ότι υπάρχουν και πολύ πάρα πολλοί ευφυείς εκτός Siemens σε πανεπιστήμια, σε ερευνητικά κέντρα και γι' αυτό είχαμε την ιδέα να συνεργαστούμε και να εργαστούμε ανοιχτά με άλλους εταίρους, ερευνητές, άλλες βιομηχανίες κλπ. Αυτό είναι αυτό που συζητάμε. Και περνώντα τώρα στο γιατί χρειαζόμαστε έρευνα στα ευρωπαϊκά προγράμματα πλαίσιο, αυτό θα είναι το δικό μου θέμα. Οι Siemens, όπως και πολλές άλλες εταιρείες, θεωρεί ότι ε, ερευνούν ε, μέσα στα πλαίσια του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του προγράμματος πλαισίου, για να βρει τους σωστούς εταίρους. Αν δεν υπάρχει σωστή χρηματοδότηση, βέβαια, κανένας δεν θα πληρώσει για το γενικό κόστος. Γιατί τον εργάζεται κανένας μέσα στα πλαίσια του ευρωπαϊκού πλαισίου, δημιουργεί υψηλό γενικό κόστος. Δηλαδή αν πάρει κανένα 50% χρηματοδότηση για ένα πρόγραμμα δεν καλύπτει τα γενικά του έξοδα. Και γι' αυτό έχουμε πάντα ένα πρόβλημα με αυτό. Το άλλο είναι, είναι το πολύπλοκο. Πολύπλοκος χαρακτήρα τη έρευνα. Δημιουργήσαμε δηλαδή ένα πολύπλοκο κόσμο, αλλά θα πρέπει να εργαστούμε για να μειώσουμε την πολυπλοκότητα και να συγκεντρώσουμε την προσοχή σε συγκεκριμένα θέματα. Και προτείνω εδώ να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας σε μεγάλες προκλήσεις, όπως είπα προηγουμένως. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για εταιρείε όπως τη δική μας και για πολλά ερευνητικά κέντρα. Το άλλο τμήμα είναι ότι έχουμε πολλές, πάρα πολλές δραστηριότητες, εκ των οποίων πολλές είναι εκ παραλίλου. Θα θέλαμε λοιπόν Λιγότερε, αλλά μεγαλύτερε και πιο ισχυρέ πρωτοβουλίε. Παράδειγμα, ένα από τα θέματα που συζητάμε αυτή τη στιγμή είναι το διαδίκτυο του μέλλοντος, πάρα πολύ σημαντικό θέμα για την Ευρώπη, γιατί προφανώς το παλιό διαδίκτυο είχε οριστεί στις ΗΠΑ, το μελλοντικό όμως διαδίκτυο θα είναι ένα διαδίκτυο αγαθών, υπηρεσιών, γνώσης και αυτό μας δίνει Καινούριε ευκαιρίες. Υπάρχουν δηλαδή σημαντικές ε, αλλαγές και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ορίσουμε τον νέο κόσμο του διαδικτύου. Και νομίζω ότι το ξέρει αυτό η Κομισιόν. Υπάρχει μια ομάδα που λέγεται ΕΦΙΑ που ασχολείται με αυτό, μια που λέγεται ΦΥΡΑ για το μέλλον και τα ευρωπαϊκά τεχνολογικά προγράμματα ETP εξακολουθούν να υπάρχουν πιο γνωστά από αυτά σχετικά με το ε, μελλοντικό διαδίκτυο είναι το ΝΕΣΥ και εγώ είμαι ε, παρεμπιπτόντως και πρόεδρος ε, της ομάδας αυτής. Εδώ νομίζω χρειαζόμαστε κατεύθυνση για να δούμε πώς θα ενωθούμε, πώς θα συνεργαστούμε οι οργανώσει και οι εταιρείε που υποστηρίζουν αυτέ τι δραστηριότητε, εκ των οποίων οι περισσότερε υποστηρίζουν πάνω από μία, ενδιαφέρονται να υπάρχει καλύτερη εστίαση και όχι τόσο πολύπλοκα προγράμματα. Το άλλο θέμα που ήθελα να σα πω είναι η γλυγορότερη λήψη αποφάσεων και εφαρμογή. Δηλαδή, σήμερα που όλα περνάνε από το διαδικτύο, η ταχύτητα έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία. Σε ορισμένε περιπτώσει είμαστε πολύ γρήγοροι, αλλά όχι επαρκώ γρήγοροι. Ένα παράδειγμα το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογία Πρώτη συζήτηση με τον πρόεδρο Μπαρόζο το 2006 και το, η πρώτη εφαρμογή των πρώτων κέντρων έγινε το 2010-2011. Ε, τώρα ξεκινά προς... Έχουμε κατόπιν να αρχίσουμε να εργαζόμαστε πραγματικά. Ταυτόχρονα όμως είχαμε το Facebook, την εισαγωγή του iPhone και iPad από το Apple και η η Siemens που ξεκίνησε με 800 άτομα μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και τώρα έχει φτάσει από τους 80 στους 1000. Γιατί αν δεν περάσουμε γλίγορα από την απόφαση στην εφαρμογή, ίσως δεν υπάρχει τίποτα πια ενδιαφέρον να εφαρμοστεί. Ο συσχετισμός αυτός μεταξύ της, του συσχετισμού των ευρωτικών επιχειρήσεων με την παιδεία, με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, εξακολουθεί να παραμένει. Τώρα που θα ήθελα να αναφέρω, έχω την εντύπωση ότι όσο πάει περνάμε σε ένα σκεπτικό ελέγχου, δηλαδή δεν βασίζεται στην εμπιστοσύνη η έρευνα και θα πρέπει στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή όταν θα δαπανούμε ένα ευρώ στην ε, καινοτομία αυτή καθημερινή, καταβούμε άλλο ένα στους ελέγχους, στις αιτήσει, στις παρουσιάσεις κλπ. Αυτή η σχέση όμως δεν είναι σωστή, γιατί αν έχουμε καλύτερη βάση εμπιστοσύνη, αν ε, έχουμε εμπιστοσύνη δηλαδή σε αυτούς οι οποίοι επιδίνουν τα χρήματά τους, άμα μιλάμε για βιομηχανικές εταιρείες, θα μειώσουμε το κόστος και τις προσπάθειες. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνεται ένα έλεγχο εκ των υστέρων, αλλά το θέμα είναι τι σχέσει μεταξύ τη δαπάνη για την ε, καινοτομία και τη δαπάνη για του ελέγχου. που θα πρέπει να είναι καλύτερη ισορροπημένη νομίζω. Έρχεται κλειδί. βρισκόμαστε στη σωστή άγουσα, αλλά θα πρέπει να νιώσουμε την πολυπλοκότητα, να καθορίσουμε τι προτεραιότητε να δράσουμε γλυγορότερα να αποφασίζουμε σύμφωνα με την απόδοση και να εργαστούμε με βάση την εμπιστοσύνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρος. Πάρα πολύ ενδιαφέρον οι πληροφορίε που μα δώσετε κι εσεί και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον Μαρκ Σουμπλά, <coughs> Σουμπλίν Σουμπλά, που είναι Head of Management Management Product Development European Investment Fund. Παρακαλώ. Thank um, um, Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Και είμαι ευτυχής που έχω την ευκαιρία να συμβάλλω στην εργασία σας και να απαντήσω και στις ερωτήσεις σας. Επειδή είμαι πολύ πειθαρχημένος, ακολούθησα τις υποδείξεις της γραμματείας και θα κάνω την παρουσίασή μου στην ε, μετρική μου γλώσσα. Ο στόχος της παρουσίασης αυτής θα είναι να σας ε, ενημερώσω για την εμπειρία μου όσον αφορά τη διαχείριση του προγράμματος ε, καινοτομίας και να ε, καταλήξω σε κάποια διδάγματα και να σας δώσω ίσως και κάποιες θετικές συμβολές. Στη χώρα μου είμαστε το, το τμήμα της ομάδας ΕΜΠΕΙ που ασχολείται με την εγγύηση και τη διαχείριση του κεφαλαίου και ακολουθούμε όλη την αλυσίδα ε, της ε, των επενδύσεων. Διαχειριζόμαστε πόρους στους οποίους μας, μας εμπιστεύεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης τα κρατημέλη στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής. Θα σας παρουσιάσω βασικά τις δραστηριότητές μας στα επισφαλή κεφάλαια και στις εγγύησεις και στη συνέχεια θα δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα εν ώψη των μελλοντικών προγραμμάτων. Το και επισφαλή κεφάλαια είναι βασική, βασική δραστηριότητα. Είναι μια κυκλική αγορά που πρόσφατα γνώρισε πολύ έντονες κρίσεις το 2000 και το 2008 και τα ποσά των κονδυλίων που συγκεντρώθηκαν το 2010 έφτασαν μόνο τα 2 δις ευρώ από τα οποία, δηλαδή τουλάχιστον εν τρίτο των ε, δημοσίων κονδυλίων χάρη στους επενδυτές, η αποδοτικότητα του τομέα είναι αδύναμη και αρνητική και υπάρχει πολύ μικρή έξοδο στο χρηματιστήριο, η αγορά είναι μπλοκαρισμένη. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια πως οι τεχνολογικές επιχειρήσεις που είναι υποψήφιες για χρηματοδότηση από επισφαλή κεφάλαια γιατί δεν μπορούν να πάρουν ε, τραπεζικά δάνεια έχουν εξαφανιστεί. Όχι, η τεχνολογική βάση εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά υπάρχει θέμα χρηματοδότησης. Και ιδιωτική χρηματοδότηση πιο συγκεκριμένα. Γι' αυτό πρέπει να χρηματοδοτηθεί αυτό ο τομέα. Εδώ και 10-12 χρόνια που δρούμε στον τομέα έχουμε χρηματοδοτήσει πάνω από 350 ε, ταμεία επισφαλών κινδύνων. Ε, προσπαθούμε να προσελκύσουμε ιδιωτικό κεφάλαιο. 5 δις ευρώ για λογαριασμό της ε, ΕΤΕ έχουμε διοχετεύσει και είμαστε υπεύθυνοι για το early stage, δηλαδή στην την αρχική φάση, το κεφάλαιο κίνησης στην Ευρώπη. Η παρέμβασή μας μπορεί να φτάσει μέχρι το 50% του μεγέθους των κονδυλίων όπου επενδύουμε. Είμαστε ως επενδυτής ε, ως δημόσιος δηλαδή οργανισμός που εξαρτάται από την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί βασικός μας μέτοχος είναι η ΕΤΕ και η Κομισιόν είναι ο άλλος μας μέτοχος είμαστε πολύ βασικοί για την επιβίωση της αγοράς. Τι προσπαθήσαμε λοιπόν να κάνουμε μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε και να μεταβάλουμε το πρότυπο παρέμβασης. Κλασικό μοντέλο ήταν η παρέμβαση στα κονδύλια. Αλλά έπρεπε και τα κονδύλια να μπορέσουν να ξεκινήσουν. Έπρεπε να φτάσουμε μέχρι 50% αρχικά και είχαμε μέχρι 50% γιατί το άλλο 50% ήταν ιδιωτικά κονδύλια. Προσπαθήσαμε λοιπόν με ιδιωτικά κονδύλια να διευκολύνουμε σύγχρηματοδότηση, επενδύσεις κοινέ στη Γερμανία, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία στο Ηνωμένο Βασίλειο, UKFTF, με δημόσιους οργανισμούς για να χρηματοδοτήσουμε την τεχνολογία στις χώρες αυτές. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να αναπτύξουμε το corporate venturing, όλο ένα και περισσότερο με μεγάλους τέρους της βιομηχανίας, ε, με φαρμακοβιομηχανίες συνεργαζόμαστε και ελπίζουμε να συνεργαστούμε και με επιχειρήσεις ε, του τομέα της ε, πληροφορικής. Ε, δουλεύουμε λοιπόν και συνεργαζόμαστε στενά με εθνικούς εταίρους αυτή τη στιγμή ίσως να το είδατε και στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναζητούμε, προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα ταμείο για τις ευρεσιτεχνίες και την πνευματική διοκτησία σε συνεργασία με το ΚΕΣΕΝΤ με διάφορες ε, αντίστοιχες οργανισμούς στη Γαλλία, Ιταλία και αλλού. Έχουμε αναπτύξει όλο ένα και περισσότερο την δραστηριότητα της μεταφοράς τεχνολογίας, ευνοώντας τη σύνδεση ανάμεσα στα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα και την αγορά. Προσπαθήσαμε δηλαδή να βρούμε νέους δρόμους και στο μέλλον θα πρέπει να αναπτυχθούν περισσότερο, να έχουμε αρκετά ευέλικτα μέσα ώστε να προχωρούμε διαρκώς και να, να ζητούμε νέες κατευθύνσεις για να διευκολύνουμε τις δράσεις μας. Ήθελα να σας δώσω ένα παράδειγμα για την ανάπτυξη της δραστηριότητας για την μεταφορά των τεχνολογιών που αφορά για παράδειγμα την ανάπτυξη των μικρών επιχειρήσεων, το spin-out, ε, δραστηριότητες ε, διοδότηση ή συμφωνίες συνεργασίας το πρόγραμμα που έχουμε αυτή τη στιγμή, το οποίο περιορίζεται στι μικρομεσαίες επιχειρήσει, δεν μα επιτρέπει, για παράδειγμα, να χρηματοδοτήσουμε τέτοιου είδους δράσεις, γιατί η αδειοδότηση που χρηματοδοτούμε συνήθω χαίρει, μάλλον ωφελεί μεγάλε επιχειρήσει και άρα δεν είναι επιλέξιμο. Είναι ένα θέμα στο οποίο θα επανέλθω όσον αφορά το συμπέρασμα στο οποίο μπορούμε να καταλέξουμε. Όμω, είναι ένα τομέα όπου πρέπει να βρεθούν κονδύλια και να βοηθήσουμε να δημιουργηθούν οι χρηματοπιστωτικές αυτές δομές ώστε να ευνοηθεί η σύνδεση ανάμεσα στα ερευνητικά κέντρα και την αγορά. Στο UMIC, το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, χρηματοδοτήσαμε το τελευταίο ε, βραβείο Νόμπελ, τον καθηγητή Βόσελοφ, που με τα νέα υλικά που ανέπτυξε ε, χρηματοδότησε χρηματοδοτήθηκε μάλλον από αυτό το πανεπιστήμιο και από αυτό το κονδύλι. Τώρα, στην περίπτωση του ΣΥΠ που θα ολοκληρωθεί το 2013, έχουμε υπογράψει για 220 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι δηλαδή κάλυψη κινδύνου, εγγύησεις που επιτρέπουν να καλυφθεί ο κίνδυνος για πάνω από 3,8 δις για μικρομεσαίες, για δάνεια σε μικρομεσαίες. Αφού του είδους η δράση λοιπόν έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο μόχλευσης, ε, βελτιώνει την δημόσια ευαισθητοποίηση, είναι ένας τομέας πολύ σημαντικός συνεργασίας με τους εθνικούς εταίρους. Από τις 80.000 επιχειρήσεις που έχουμε χρηματοδοτήσει στο πλαίσιο του ΣΥΠ, θεωρούμε πως το 50% είναι επιχειρήσεις καινοτόμες. Και θα πρέπει να σας πω ότι μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία της τάξης του 80% ήταν επιχειρήσεις με λιγότερο από 10 ε, ε, υπαλλήλους. Μικρές επιχειρήσεις, όχι συστηματικά καινοτόμα με την ε, Γενική Διεύθυνση Έρευνα και την ΕΤΕ προσπαθούμε να δούμε πώ θα φτιάξουμε για το 2012 και 2013 μία πτυχή μικρομεσαίε για την ε, ε, δυνατότητα εξέβρεσης κοινού επισφαλούς κεφαλαίου έχει λειτουργήσει για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Όμως θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι αντίθετα με την δραστηριότητα SIP, που γενικά είναι στοχευμένη για τις καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, α, συγγνώμη, που είναι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τις καινοτόμε επιχειρήσεις είναι πολύ πιο δύσκολο να εφαρμοστεί, γιατί οι τράπεζες έχουν γενικές δραστηριότητες, έχουν ένα χαρτοφυλάκι για τις μικρομεσαίες. Τίθεται το θέμα της επιλογής των καινοτόμων επιχειρήσεων. Άρα λοιπόν θα πρέπει να πάμε να βρούμε στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών με τι οποίε έχουμε συμφωνίε. 10, 20, 15, 500 μικρομεσαίες που θεωρούνται καινοτόμες και τις οποίες θα βάλουμε σε ένα σύνολο και τις οποίες, για τις οποίες θα αγγιηθούμε και θα κάνουμε συμφωνία με 30-40 τράπεζες. Αλλά πάντως πρέπει να βρούμε τις επιχειρήσεις στις τράπεζες και να τις συγκεντρώσουμε και να αγγιηθούμε για αυτές. Είναι περίπλοκο να γίνει κάτι τέτοιο. Πρέπει να έχει μια σχέση πολύ προωθημένη με τις τράπεζες και τίθεται και το πρόβλημα, αν μιλάμε για κρατικά χρήματα, επιλεξιμότητας. Δηλαδή, πρέπει πολύ σαφώς να υπάρχει συμφωνία για τον ορισμό της καινοτομία. Σε περίπτωση δηλαδή ελέγχου, ελεγκτικό συνέδριο, αν τα κριτήρια δεν είναι σαφή, αν δεν μπορούν να τηρηθούν, οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να αποζημιώσουν για κονδύλια. Πράγμα που έχει τελείω αρνητικό αποτέλεσμα για την εφαρμογή όλη αυτή τη διαδικασία. Η σαφήνεια της του ορισμού για την καινοτομία είναι πολύ σημαντική. Αλλά είναι αλήθεια ότι γνωρίζουμε πως δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτή την στοχευμένη εγγύηση για τις επιχειρήσεις, είτε είναι καινοτόμες είτε όχι, είτε είναι σε άλλους τομείς για την επάρκεια σε ενέργεια, περιβάλλον ή άλλους τομείς. Μπορεί να είναι και η βιομηχανία ε, του πολιτισμού που, είναι, που έχουν καινοτόμο χαρακτήρα και είναι στατική σημασία για την Ένωση. Κάποια διδάγματα που μπορούμε να αποκομίσουμε από τη δραστηριότητά μας και σημεία για τα οποία θα ήθελα κάπως να επιμείνω. Απαραίτητη προσθέμενη αξία ενό καινοτόμου προγράμματο εξαρτάται από την γεωγραφική του θέση, από τις σύνθηκες της αγοράς και δεν μπορεί να αποφασιστεί εκ των προτέρων. Το να πούμε για παράδειγμα ότι ένα παράδειγμα αυτομάτως θα πρέπει να αφορά προγράμματα ή κονδύλια διαμεθοριακά είναι ε, παρακινδυνευμένο. Στο θέμα των επισφαλών ε, κεφαλαίων. Αν πάμε ας πούμε, σε ένα νέο κράτος μέλος όπου δεν υπάρχουν επισφαλή κεφάλαια και όπου θα φτιάξουμε ένα κονδύλιο για, ένα αναπτυξη... για αναπτυξιακά κεφάλαια θα ήταν επιτυχία. Ε, είναι ήδη επιτυχία στη Γαλλία ή στην Αγγλία όπου η αγορά είναι πιο ανεπτυγμένη. Εκεί τα ευρωπαϊκά χρήματα πρέπει να μπουν πολύ πιο νωρί ε, στο στόχο, δηλαδή στην επόαση, στην ε, εκτίμηση, στην τιμολόγηση και ούτω καθεξής. Και αυτή η προστιθέμενη αξία μεταβάλλεται με τον χρόνο. Όταν το 98-2000 η αγορά των επισφαλών κεφαλαίων μπορούσε να συγκεντρώσει 20 δις ευρώ από ιδιώτες, τα δημόσια χρήματα τότε έπρεπε να πάνε πολύ πολύ πιο μπροστά στον κύκλο. Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο μόλις δις. Όπω καταλαβαίνετε αυτό εξαρτά, ε, ε, επεκτείνεται σε ολόκληρη την αγορά. Είναι θέμα επιβίωσης. Αν σε τρία χρόνια ανεβεί πάλι η αγορά, φυσικά η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία θα πρέπει και πάλι να προσαρμοστεί αναλόγω. Υπάρχει μια ανάγκη λοιπόν για μόνιμη παρακολούθηση των συνθήκων της αγοράς για να βελτιστοποιηθεί η χρήση των κονδυλίων και αυτό ισχύει και για τις εγγύησεις εξάλλου. Το δεύτερο επί το οποίο θα ήθελα να επιμείνω είναι η επικουρικότητα, η ανάγκη να συνεργαστούμε στενά με εθνικούς εταίρους ώστε να τους επιτρέψουμε να κάνουν περισσότερα και καλύτερα και σε κάποιους τομείς και θα σας μιλήσω σύντομα για το Ταμείο Ευρεσιτεχνιών το οποίο μελετούμε αυτή τη στιγμή με εταίρους όπως η ΚΕΣ η ΚΑΒΕ, η ΚΑΖΑ ο τομέας της πνευματικής ιδιοκτησίας, ε, του Ταμείου ε, για τις ευρεσιτεχνίες, όπως έχουν φτιάξει οι Ιάπωνες και φτιάχνουν και οι Αμερικάνοι. πρέπει να συγκεντρώσει προσπάθειες και των εθνικών εταίρων. Έπειτα, επενδυτικές κατευθυντήριες γραμμές και αυτές θα πρέπει να τις ε, φτιάξουμε θα ήταν αλαζονικό να, να πιστεύουμε ότι μπορούμε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες της αγοράς ή όλα τα κενά της αγοράς για μια τόσο μακρά περίοδο, μια δεκαετία. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για αυτές τις κατευθύνσεις γραμμές και λέμε ότι πρέπει να αυτές να ισχύουν για δέκα χρόνια. Όμως πρέπει να έχει κανείς μια βάση νομική σύντομη που επιτρέπει να διολυσταίνουν οι δράσεις ανάλογα με τις ανάγκες αυτή την έλλειψη ευελιξία την αισθανθήκαμε όταν χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε την κρίση και είδαμε ότι οι κατευθύνε γραμμές που είχαμε που έπρεπε να εφαρμόσουμε είχαν καθοριστεί για μια περίοδο που δεν ήταν περίοδος κρίσης και μας ενοχλούσαν. Δεν μπορούσαμε να αντιδράσουμε όπως θέλαμε. Τέλος, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια εικόνα που θα βασίζεται στη συμπληρωματικότητα και τη σωστή διάρθρωση ανάμεσα σε όλες τις ενέργειες, σε όλες τις δράσεις που γίνονται για την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Το πρόγραμμα για την καινοτομία, το πρώην ΣΥΠ, υπάρχουν διάφορες ενέργειες δράσεις από το Διευθυντικό Ταμείο. Διαχειριζόμαστε και το ΦΕΝΤΕΡ, όπου φτιάχνουμε και εκεί εγγυήσει και επισφαλή κεφάλαια με τα εθνικά χαρτοφυλάκια. Υπάρχουν ε, τα δάνεια της ΕΤΕ, επιδοτήσεις, οι δράσεις των εθνικών ε, ε, θεσμών, η ανάγκη για τεχνική βαρογή. Όλοι αυτοί οι φορείς θα πρέπει να συντονιστούν με τρόπο θεσμοθετημένο σχεδόν για να δούμε πώς μπορούν να βελτιστοποιηθούν οι δράσεις τους ανά περιοχή, ανά ζώνη με τακτικό τρόπο γιατί διαφορετικά θα γίνουν επικαλύψεις οι οποίες έχουν αρνητικές επιπτώσεις. Αυτά τα βασικά που ήθελα να σας αναφέρω. Στόχοι που εμείς βλέπουμε είναι οι στόχοι επί των οποίων ήδη δουλεύουμε, δηλαδή μεταφορά τεχνολογίας, σύνδεση ανάμεσα στα κυβερνητικά κέντρα και την αγορά, την ε, πνευματική διοκτησία, υποστήριξη στους business angels που είναι διστακτική σε κάθε δομή αλλά που αποτελούν ένα μεγάλο κομμάτι του κεφαλαίου εκκίνησης, ε, τα ταμεία των επισφαλών κεφαλαίων, και στο θέμα της καινοτομίας να έχουμε έναν ορισμό αρκετά ευρύ ώστε να καλύπτει και τομείς όπως ας πούμε η κοινωνική καινοτομία. Εμείς επιθυμούμε να παίζουμε πρωτοπόρο ρόλο, και κλικό σε σχέση με την αγορά. Αυτός είναι ο ρόλος ενός κρατικού φορέα και δημόσιο φορέα υπέρ των ΜΕ και να καλύψουμε και άλλες επιχειρήσεις που είναι σε ανάπτυξη και που κάποιες φορές ξεπερνούν πια το στάδιο της μικρομεσαίας. Σα μίλησα για οικονομικά θέματα και χρηματοπιστωτικά μέσα. Υπάρχει ένα πλαίσιο που είναι απαραίτητο για την εφαρμογή αυτών των μέσων. Είναι το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνία. Είναι μια φορολογική μεταρρύθμιση που θα εμποδίζει τη διπλή φορολόγηση. Μεταξύ άλλων, μεταξύ άλλων, αλλά που είναι στοιχεία ε, απαραίτητα σε συνδυασμό με τα δημοσιονομικά μέσα. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Εμείς ευχαριστούμε. Πάρα πολύ δύσκολα είναι όλα αυτά, περίπλοκα. Για να μπορούν να έχουν περισσότερη καινοτομία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Σας ευχαριστώ. Χρειάζομαι ορισμένα δευτερόλεπτα, γι' αυτό έτσι μακρηγορώ. Γιατί πρέπει να ξαναξεκινήσει το μηχάνημα με την επόμενη ομιλία. Χρειαζόμαστε δύο-τρία λεπτά. Και θα περάσουμε με τον επόμενο εισηγητή. Και τηρούμε πολύ καλά τον χρόνο μας, γιατί όλοι πραγματικά προσπάθησαν όλοι οι επισκέπτες μας και το κατάφεραν κιόλα να είναι πιο σύντομοι. Και αυτό δεν είναι μια τεράστια ευκαιρία να έχουμε πολλές ερωτήσεις και πολλές ευφύες απαντήσεις βέβαια. Εντάξει? Mm. Όχι, ακόμα λεπτό. Λοιπόν, ο επόμενος που θα πάρει το λόγο θα είναι ο κύριος Βαζάρα. Head of Global Consulting Practice in Innovation από τη Φιλανδία. Σας καλωσορίζω κύριε Βασάρα. Νομίζω ότι μπορείτε να πάρετε το λόγο τώρα, να μας κάνετε την παρουσίασή σας. Σε μερικά δευτερόλεπτα είναι έτοιμο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. So, thank you. Σας ευχαριστώ πρώτα πρώτα που με καλέσατε. Σε αυτήν σημαντική εκδήλωση Βέβαια, το, η υπηρεσία μας ε, έχει ένα όνομα πολύπλοκο. Όνομα πολύπλοκο δύσκολο και να το προφέρει κανείς, αλλά τέλος πάντων ασχολούμαστε στη, με αυτή την υπηρεσία στη Φιλανδία εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ε, πάντως ε, άλλο το τι κάνουμε εμείς, άλλο το τι κάνετε εσείς. Δεν θα σας πω ότι πρέπει να μας μιμηθείτε όμως, να σας πούμε ποια είναι η δική μας ερμηνεία των πραγμάτων. Πρώτα-πρώτα αποτελεσματικότητα της χρήσης των πόρων. Έχουμε Είμαστε 5 εκατομμύρια, ζούμε στο βορρά, βιομάζα, επομένως και εγκέφαλος και ξυπνά δεν χρειάζεται και πρέπει να τα χρησιμοποιεί κανείς αποτελεσματικά. Τώρα έχουμε αυτό, τη δική μας εκδοχή της καινοτομία. Έχουμε εταιρείε ερευνητικές που δρούν σε θύλακες κατά το ίμιση για την ερευνητική δραστηριότητα χρηματοδοτεί το κράτος για αυτό το σοξ όπως το λέμε είναι, ε, η δράση έχει χτυπηθεί φυσικά για την ύφεση και έχουμε ε, πάρα πολλές θεωρίες για το, για το πώς εξελίσσεται η ύφεση, αν έχει το σχήμα του L, του λατινικού, του U, του V, του W. Όμως εμείς λέμε ότι φταίει κάτι άλλο, φταίει η ασυνέχεια. Η ασυνέχεια είναι μεγάλο πρόβλημα. Ιδίω όταν κανείς δεν μπορεί να κάνει τη διαφορά. Άρα να δούμε πώς μπορεί κανείς να προστατευτεί από αυτή την ύφεση, ε, να δει κανείς, τι μπορεί να κάνει από, από τις... Ε, διαδοχικές συνεχιζόμενες υφέσεις. Ξέρω όλα αυτά είναι σε κλασικές συμβουλές εταιρεία συμβούλων, αλλά θέλω να σας δώσω αυτό το μήνυμα και έχουμε εδώ πέρα ε, τρία πράγματα τα οποία έχουν στα, στα αγγλικά αρχικό το D, Είπαμε ότι θα πρέπει να μην υπάρχει κατάσταση της αγοράς, θα πρέπει να υπάρχει απορρίθμιση και θα πρέπει κανείς να αμήνεται όταν ο χώρος του υφισταται επίθεση. Είπαμε όχι επίσης ε, εάν κανείς ε, είναι κάπου ισχυρό, θα πρέπει να ενισχύεται περισσότερο Είμαστε πρωτοπόροι για την καινοτομία σε όλο τον κόσμο, αλλά ταυτόχρονα ε, μας λείπουν κάποια μέταλλα, άρα η χημική βιομηχανία είναι πρωτοπόρα, αλλά θα πρέπει να βρει τρόπο να παραγάγει αυτά τα μέταλλα που λείπουν. Αυτά όσον αφορά την κινητικότητα. Δεύτερον, ε, περιέργεια, ερευνητικό πνεύμα, Είμαστε πολύ πιο προχωρημένοι στα επιστημονικά ζητήματα πόσο σκέφτεστε περισσότερο από εσά. Θέλουμε να ξέρουμε τι γίνεται, θέλουμε να είμαστε πρωτοπόροι και επομένως για τους άλλους λέμε ότι αντί να μας αντιγράφουν θα πρέπει να τους αντιγράφουν. αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε ότι έχουμε τα, τα, τα μυαλά αλλά δεν έχουμε την αντίστοιχη οργάνωση. Υπάρχει το θέμα βεβαίως της ευρωπαϊκής αδειοδότησης. Δεν μπορούμε να ξαναφέρουμε τον τροχό, δεν είμαστε τόσο έξυπνοι. Απλώς αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να, τον τροχό να τον αξιοποιήσουμε στα πλαίσια κάποιες κατασκευές που κάνουμε επομένω, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε ας πούμε είδατε τι κάνει ο Bill Gates σε σχέση με τις επιθωτήσεις και τις εγκρίσεις είναι αυτές οι χώρες αυτές οι εταιρείε μόνο σαν του Bill Gates ε, είναι επικίνδυνε γιατί είναι φρένο στην ε, καινοτομία άρα στρατηγική που σχέση με τις ε, αδειοδοτήσεις χρειάζεται Τώρα όσον αφορά ε, την, την ε, διαίρεση, την, την πολυδιάσπαση της αγοράς, είπαμε, έχουμε εδώ ένα σωρό αρχικά τα οποία σχετίζονται με την κατάσταση της αγοράς, και λοιπά. Όμως, για να δούμε πώς είναι το τοπίο το ερευνητικό στην ε, Ευρώπη. Με σίγουρος ότι πολλοί ξέρουν, αλλά όσο περισσότερο ενοποιούμε τόσο δεν μπορούμε να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας σε ό,τι κάνουμε. Μας αρέσει αυτό το να δουλεύουμε σε ε, μικρές ομάδες, σε μικρούς θύλακες. Είμαστε μικρή χώρα άλλωστε. Και αυτό φορά και το λογισμικό. και έτσι αυτοί που εργάζονται εκεί πέρα γνωρίζουν ένα τον άλλον. Αλλά το θέμα είναι ο συντονισμός, η επικοινωνία. Αλλά έτσι πάλι ο, κάθε φύλακας σκέφτεται χωριστά. Θέλουμε πώς θα ενοποιηθεί αυτό και στην επόμενη γενιά θα είναι τα πράγματα χειρότερα. οι ερευνητές χώρου ιατρικής, ας πούμε, βιολογίας. Πρέπει να συνεργάζονται, να βλέπουν τι γίνεται όσον αφορά τη χημική βιομηχανία ουσιών που μπορούν να βγουν από ένα δάσο. Δεν μπορώ να σας πω τι έχουμε κάνει εκεί. Όμως, ακριβώς, η θεωρία λέει ότι έτσι θα πρέπει να, να γίνει και αποδίδει. Το και το πρόβλημα για μας, όπως και για όλους, είναι ότι κανείς δεν έχει παράδοση σε αυτό τον τομέα. Άρα δεν υπάρχει παρελθόν, δεν υπάρχει προηγούμενο. Όμως νερό, βιομάζα, μέταλλα και ενέργεια είναι η πόλη πρώτες που χρησιμοποιούμε και χρειάζεται όμως μια πολιτική που να ρυθμίζει όλες αυτές τις πρώτες σύλλογες τους φυσικούς πόρους χρειάζεται μια τέτοια πολιτική χρειάζεται ρύθμιση βιομάζα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα πάντα σε αυτοκίνητα ε, είδη διατροφής τα πάντα τώρα όσον αφορά την απορρίθμιση η ερώτηση είναι η εξής διαπιστώνουμε σήμερα ότι Υπάρχει ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό το οποίο θα πρέπει να επιληθεί. Έχει κάνει την ευφία, έχει ερευνητικέ ομάδες στην Ευρώπη, αλλά θεωρητικά έχει και τα χρήματα. Είναι δυνατόν όμως να έχουμε έργα, προγράμματα σε μικρογραφία του Μανχάταν, λέει ο μιλητής. γίνεται κάτι τέτοιο. Αυτό είναι που προσπάθησαν να κάνουν και το κάνανε από τη δεκαετία του 60 και μετά. Αυτό μας λείπει τώρα όσον αφορά τους εύστοχους στόχους, τους ευφύς στόχου. στόχους. Θα πρέπει να είμαστε προσαρμοστικοί. Ε, θα πρέπει να είμαστε ευέλικτοι, να αλλάξουμε κατεύθυνση αν κάτι δεν πάει καλά. Πάντως ε, έχω δουλέψει και σε αυτό που λέμε κοιλάδες. Ε, γύρω για αυτές τις κοιλάδες υπάρχουν απότομες πλαγιές όμως. Δύσκολο να τις καρφαλώσει κανείς. Και θα πρέπει επομένω κανεί να είναι κοντά μου στα διεθνή πρότυπα και θα πρέπει κανεί να τι ε, ενώσει αυτέ τι ε, απομονωμένε κοιλάδε. Και αυτό θα είναι ένα πλεονέκτημα. Επομένω χρειάζεται ελευθερία για καινοτομία, θα χρειάζεται, χρειάζεται ευελιξία και χρειάζεται και χρηματοδότηση. Βλέπετε αυτά τα τρία D που σα είπα Herzlichen Dank. Ähm, Der Kommentar, der war der Applaus. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Burton Lee, Lecturer European Entrepreneurship and Innovation. Δίνω την το λόγο στον επόμενο, στον Δ. Μπάρτον Λί, από το Stanford School of Engineering. Ήθελα να του δώσω το λόγο παρακαλώντας να μας παρουσιάσει την ομιλία του. Είναι μεγάλη μου τιμή που μπορώ να μιλήσω εδώ, που με καλέσατε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σας ευχαριστώ που έχει τη δυνατότητα το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ να κάνει μια μικρή παρουσίαση εδώ μετά που τα είπα αυτά στα γερμανικά, θα σας πω τα υπόλοιπα στα αγγλικά. Λοιπόν, θα σας πω δύο λόγια όσον αφορά τις πρακτικές για μια Silicon Valley και ειδικά ε, σχόλια για την εμπορία της έρευνας εδώ στην Ευρώπη. Είμαι αυτήν την εβδομάδα ε, σήμερα σαν εμπειρογνώμονας για το 7ο ε, προγραμμα πλαίσιο που αναθεωρούμε κάποιες προτάσεις. Θα ξαναπάω εκεί. Έχω λοιπόν κάποια εικόνα της ευρωπαϊκής σκηνής για την έρευνα και ανατομία. Ήμουνα στο Ιρλανδικό, στην Ιρλανδική Ομάδα για Καινοτομία, στη Δανία επίσης, στην Εθνική Πολιτική Καινοτομία. Συνεργάστηκα με τις ε, περιφέρειες στην Ευρώπη όσον αφορά την περιφερειακή καινοτομική ε, πολιτική, Εθνικό Σύστημα Έρευνας, ε, Εθνικό Ίδρυμα Υγεία το 2008. Είμαι επικεφαλής μια προγράμματος στο Stanford University Διδάσκω επίσης κάθε Δευτέρα. Την επόμενη Δευτέρα θα έχουμε δύο ε, καθηγητές από την Ιταλία και από την Τσεχία όσον αφορά το θέμα της ε, και της μεταφοράς της καινοτομία στην Ευρώπη. Αυτή είναι η εταιρεία που είχαμε στην Ευρώπη τα τελευταία τρία χρόνια και χώρες που, από τις οποίες έχουμε καλέσει ε, βλέπετε Εστονία, Ιρλανδία σε πράσινο αλλά και επίσης περιφερειακή, Μπαδρίτη, από την Λιό επίσης και εταιρείε ω εταίρου από την Ιταλία και αν την στην Δανία επίσης και οι πολύχρωμες χώρες είναι χώρες στις οποίες έχουμε κάτι παρουσιάσει επιχειρηματίας, τους λεγόμενους άγγελους ή έχουμε εμπειρογνώμονες. Και έχουμε επίσης ε, εκπροσώπους από την Γενική Διεύθυνση ε, των επιχειρήσεων που έρχονται στο Στάλφορ και μας μιλάνε. Θα σας πω λοιπόν τώρα για τις καινοτομίες στην ε, Silicon Valley, αν δεν την ξέρετε, είναι μεγάλη περιοχή. Λίγους κατοίκους, κάτι κάτω από 3 εκατομμύρια αλλά όσον αφορά το κεφάλαιο κινδύνου και τις επενδύσεις και υψηλή τεχνολογία, έχουμε το 40% όλου του κεφαλαίου κινδύνου που επενδύεται στις ΗΠΑ. Στον τομέα της ψηλής τεχνολογίας, ιατρική, ενέργεια, πληροφορική κλπ. Η Silicon Valley είναι το παγκόσμιο κέντρο καινοτομία σε όλο τον κόσμο, διαφορε ιδέε, τεχνολογίες, αλλά ιδίω γλίγορη μεταφορά των τεχνολογιών και των επιχειρήσεων σε διεθνές επίπεδο. Όλοι όσοι ενδιαφέρονται για τη δημιουργία των δικών τους κοιλάδων, αν θέλετε, έρχονται σε εμά για να μάθουν ε, για νέα μοντέλα, νέες τεχνολογίες, νέες ιδέες και κάποια στιγμή φτάνουν στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ για να δει πώς προχωράμε εμείς. Έχουμε συνεχίσει δηλαδή αιτήσει ε, για ε, επισκέψεις από την Ευρώπη, από τις άλλες ε, χώρες της Νοτιοαμερικής, ε, από την Ασία. Είχαμε πάρει την την περασμένο μήνα μία συνάντηση για εκπροσώπους του από τη Σανγκάη τι κάνουμε. Εμείς ε, κατασκευάζουμε εταιρείε πιο γλυγορα και πιο αποτελεσματικά από οτιδήποτε άλλο στον κόσμο. Δημιουργούμε πιο γλίγορα νέες θέσεις απασχόλησης και βιομηχανίες. Κοιτάμε ποιε είναι οι καινούριε ιδέε, τεχνολογίε και η πνευματική διακρισία που μπορεί να περάσει σε διεθνέ επίπεδο. Και επίση κάνουμε έρευνα ε, και ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο. Ιδίως προσπαθούμε μια συνεργασία από την Ιαπωνία και από την Ευρώπη φυσικά. Λοιπόν, από την κοιλάδα της Σιλικόνης, στη Silicon Valley, βλέπουμε ότι θα μπορούσε να είναι μια στρατηγική περιφέρεια για την Ευρώπη, σαν ένα τμήμα του ευρωπαϊκού καιροτοπικού οικοσυστήματος που δεν είναι καλά γνωστή στις ευρωπαϊκές ε, πρωτεύουσες. Υπάρχουν ε, πολλοί ε, εκεί Γερμανοί, Γάλλοι, Ισπανοί, Βέλγοι, Φιλανδοί, Φιλανδοί είναι πάρα πολλοί, οι Δανείοι, οι Νορβηγοί, οι Σουηδοί, οι Εστονοί. Είναι μεγάλο κέντρο δηλαδή <clears throat> επίσης ευρωπαϊκών ε, κρατικών ε, επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων από πάρα πολλές χώρες και όσο πάει υπάρχουν μεγαλύτεροι αριθμοί Ευρωπαίων επενδυτών και εφευρητών που έρχονται στη στην ε, Silicon Valley γιατί βλέπουμε ότι δεν μπορούν να προωθήσουν τις επιχειρήσεις τους όσο να γίνεται αυτό στην Καλιφόρνια. Έχουμε πολυεθνείς ε, στις τηλεπικοινωνίες, ε, αυτοκίνητο βιομηχανία, πληροφορική, αλλά έχω την εντύπωση ότι οι περισσότερε ευρωπαϊκέ χώρε και οι περιφερειές δεν είναι αρκετά δεσμευμένε εκεί στην Silicon Valley. Δεν βλέπουμε αρκετέ εταιρείε μέσου μεγέθου που έρχονται εδώ για να δουν πώ λειτουργεί η κοιλάδα σιλικόνη. Έχουμε κάποιε συνεργασίε από το Στάνφορντ με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, αλλά αυτέ είναι παλιέ συνεργασίε. <clears throat> Τα καλύτερα σχολεία, Οξφόρδη, Κέμπρο, το Επιφελέλ, ε, από τη Γαλλία επίση, το Πτυνικό Πανεπιστήμιο του, του Μονάχου Φερρυπίν, το Πανεπιστήμιο από την Τέλφ, από την Τσάλμερ, Σουηδία. Οι σχέσει αυτέ όμω μεταξύ Στάνφορτ και Μπέρκλι με, ευρωπαϊκά πανεπιστήμια είναι στη Γερμανία, στι κάτω χώρε, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στι Σκανδιναβικέ χώρε και σπάνια βλέπουμε άλλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια να έρχονται στην ε, Silicon Valley για να δημιουργήσουν αυτή τη σχέση. Ποιε είναι οι κύριε διαφορέ μεταξύ τη ε, Silicon Valley και του Ευρωπαϊκού Κοινοτοπικού Συστήματο ή η παράδοση, η σχέση όσον αφορά το κέντρο και την αποτυχία. Εμεί ε, συγχωρούμε την αποτυχία. Συγχωρούμε την αποτυχία παρά να μην έχει καμία εμπειρία όταν υπάρχει μια χρηματοδότηση καινούργια εταιρεία. Νομικά θέματα. Πανέμψαν το θέμα της, ε, της ε, αποτυχίας οικονομικής δεν επιβαρύνει. Είμαστε ανοιχτοί όσον αφορά την, ε, ε τις κοινέ πληροφορίες, την συναλλαγή πληροφοριών, ανταλλαγή πληροφοριών. Δεν είμαστε σκεπτικές, είμαστε ε, αισιόδοξοι, έχουμε ανοιχτό δίκτυο, έχουμε διαδικασίες επιχειρηματίες που κινούνται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι στην Ευρώπη ή σε άλλο μέρος του κόσμου. Ελάχιστο ρόλο της κυβέρνησης, καμιά φορά σημαντικό όμως για την επένδυση της έρευνας, πολλά μοντέλα θεσμικά, εθνικά, startup ε, επιχειρήσεις, ε, κρατικά, μεγάλες αγορές. Όλα αυτά όσον αφορά την κρίσιμη μάζα και την κλίμακα εργασίας και επίσης πολύ ισχυρά εσωτερικά δίκτυα στην Κοιλάδα, αλλά επίσης συνεχώς νέες διασυνδέσεις εκτός της Κοιλάδας, στην Ασία, στην Ευρώπη και αλλού. Γι' αυτό τώρα αρχίζουμε να βλέπουμε από τη Βραζιλία αντιπροσωπείες να έρχονται. Η Χιλή επίσης. Κίνα, Ινδία, Σιγκαπούρη, Κορέα, εκεί πολλοί ε, φοιτητέ ε, στο Στάνφορντ, στο Μπέρκελι. Και από την Ευρώπη βέβαια, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει το επίπεδο δέσμευσης που χρειάζεται η Ευρώπη. πραγματοποίηση νέων εταιριών γιατί συγκεντρώνουμε το κεφάλαιο κινδύνου, τους, ε, την πρόσβαση στην αγορά. Οι πελάτες μας είναι εταιρείε ή καταναλωτές που είναι εκείνοι που προσαρμόζονται γλυγορά. Τυπικά έχουν πρόσβαση στην πιο πρόσφατη τεχνολογία στους περισσότερους τομείς. Ε, συλλέγουμε τους ηγέτες σκέψης ε, σε παγκόσμιο κλίμακα Πολλοί που έρχονται μένουν βέβαια στι ΗΠΑ, ορισμένοι επιστρέπουν. Έχουμε διαφορετικά <clears throat> μοντέλα καινοτομία για τα πανεπιστήμια από ότι εδώ είμαστε το επίκεντρο της καινοτομία και βέβαια λόγω της διαφορετικής μας έχουμε πολύ στενές σχέσεις με την Κίνα, τη Σιγκαπούρη και την Ιαπωνία. Εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να αυξήσει, ότι αυξάνεται μάλλον η σημασία της ε, κοιλάδας σιλικόνης για την Ευρώπη θα πρέπει να μπορεί να δουν η Σλοβακία, η Σλοβανία, τα Βαλκάνια, η Ανατολική Ευρώπη. Τώρα αρχίζει να κατανοεί ότι χρειάζεται κάτι τέτοιο. Ορισμένες από τις στάσεις που θα ήθελα να σας υποβάλω για την κοινοτική και ενατομική ε, στρατηγική να υπάρχει στενότερη σχέση με την κοιλάδα της Λικόνης, με τη Silicon η Ευρώπη δεν υπήρχε στο ίδιο επίπεδο όπω η Κίνα, η Ινδία και η Ιαπωνία όσον αφορά τη δέσμευσή τη με θεσμικά όργανα της Silicon Valley. Χάνει έδαφο η Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Συγκεκριμένα σχόλια τώρα όσον αφορά την εμπορία της έρευνας. Κατά τη γνώμη μου, μια που ήμουν σε πολλά σχέδια του δόμου προγράμματος πλαισίου της ευρωπαϊκής έρευνας δεν βλέπω να υπάρχει αρκετή σύνδεση με προϊόντα που τη χρειάζεται η Ευρώπη. Συζήθηκα, συζήτησα με πολλούς και υπάρχει νομίζω μία άποψη που προβλέπει ακαδημαϊκή έρευνα αφενός και εμπορία αφετέρου. Ότι τα δύο είναι ασύμβατα. Εμείς στο Στάντφορτ έχουμε αναπτύξει μια προσέγγιση με την οποία διατηρούμε την ακαδημική ε, πειθαρχία του Πανεπιστήμιου. Ταυτόχρονα έχουμε όμως και έντονη, έντονο προσανατολισμό στην εμπορία. Δεν λέω ότι είναι δυνατή η εμπορία κάθε προγράμματος του εβδόμου προγράμματος πλαίσιο, αλλά υπάρχουν δυνατότητες πολλές φορές που δεν χρησιμοποιούνται. Δεν ζητάτε δηλαδή από τους υποβάλλοντες συζητήσεις να συζητήσουν το θέμα του συσχετισμού μεταξύ της εμπορίας και της έρευνας που θα έπρεπε να είναι μια κεντρική ιδέα και του και νομίζω και του 8ου προγράμματος πλαίσιο. Νομίζω λοιπόν ότι τα ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να έχουν ξεκάθαρο συσχετισμό και ε, άγουσες προς την ε, εμπορία. Εδώ έχουμε λοιπόν ένα ευρύ πλαίσιο να ληφθεί υπόψη η ε, έρευνα και να προχωρήσει στην εμπορία. Ε, ε, θα πρέπει κανένας να έχει κατά νου τα κύρια βήματα της έρευνας. Εδώ στα αριστερά έχουμε την βασική έρευνα πριν από τον εγωρισμό, από το 7ο και το 8ο πρόγραμμα πλαίσιο, χρειάζεται μετά ένα ενδιάμεσο στάδιο που περνάει σε, ένα, σε μια πρώτη φάση από τα εργαστήρια και μετά περνάει στην εισαγωγή στην αγορά. Σήμερα η γραμμή μεταξύ της έρευνας και της, ε, εμπορίας η, η μετάφαση από το ένα στο άλλο δεν είναι δυνατή δεν υπάρχει εισαγωγή εταιριών προς επενδυτές που μπορούν να τους βοηθήσουν να δημιουργήσουν νέε εταιρείε, παραδείγματο χάρη. Το πρώτο βήμα είναι ένα πλαίσιο της εμπορία τη ε, έρευνα για να δουν πώς λειτουργούσε αρχικά το 7ο και το 8ο πρόγραμμα πλαίσιο και τι θα πρέπει να γίνει. Αυτά τα δύο δηλαδή αριστερά ε, δεξιά σημεία δεν έχουν εφαρμοστεί συγκεκριμένα μέτρα μπορούν να υιοθετηθούν για να προχωρήσουν ε. να υπάρχει ε, εξολόγηση των κριτηρίων και όσον αφορά τα στοιχεία που ζητούν κατά την υποβολή αιτήσεων να μπορέσει να συμπεριληφθούν το κεφάλαιο κινδύνου αυτοί οι λεγόμενοι άγγελοι, επιχειρηματίες, ε, νομίζω ότι θα υπήρχε κάποια αξία στο να είναι πιο ορατά τα αποτελέσματα του προγράμματος πλαίσιο. Να υπάρχει παραδείγματο χάρη μια τράπεζα στοιχείων όπου όλα τα ε, αποτελέσματα της έρευνας της να μπορεί να ε, ευρυθούν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό έτσι να ξέρει κανένα τι γίνεται με αυτή την πνευματική ε, ιδιοκτησία που δημιουργείται και να υπάρχει και μια ακολουθία, δηλαδή τι γίνεται, πόσε πόσες ευρυστηχνίες παρήχθησαν, τι κάνανε με τις ευρυστηχνίες αυτές και ούτω καθεξής. Βέβαια αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα ε, προγράμματα του 7ου προγράμματος πλουσίου. Ορισμένα είναι πολύ βασικής έρευνας που δεν μπορούν να περάσουν εμπορία. Ε, εμένα μου είπανε προσωπικά ε, οι υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής ότι όταν κάνω την αξιολόγηση των ε, αιτήσεων δεν θα πρέπει να λαμβάνω υπόψη το κατά πόσον έχει μια πρόταση ένα εμπορικό δυναμικό. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ μεγάλο σφάλμα. Λοιπόν, εγώ πρόκειται από την ε, αεροναυπηγική, την πολιτική και την έρευνα του διαστήματος. Αυτό που λάσαμε στιγμή είναι ότι θα υπήρχε μία ενιαία δομή για την εμπορία των ε, ε, σχέσεων με τους εμπορικούς τομείς, δηλαδή με τους λεγόμενους άγγελους επενδυτές κλπ. Για να υπάρχει παραδείγματος χάρη έτσι ένα σχετισμός από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για το διάστημα με το δίκτυο της ΕΣΑ. Ίσως κάτι μπορεί να υπάρχει εκεί, να υπάρχει εξ αυτού ένας συσχετισμός όπου οι διαδικασίες υποδομή να περάσουν κατευθείαν στα προγράμματα ΕΣΑ. Δεν θέλω να πω πολλά ακόμα. Εγώ είδα τα θέσει της EBN και της ΕΝΕΣΑ, τα σχέδια πολιτικής που υποβάλλουν στην Ευρωπαϊκή Κομισιόν. Μου φαίνεται ότι είναι καλογραμμένα και ότι λαμβάνεται πραγματικά πολύ καλές ε, συμβουλές από τις οργανώσεις αυτές αυτά. Και για να τελειώσω, ορισμένα άλλα θέματα που αξίζουν τη προσοχή, που προέρχονται από την Ελλάδα που έκανα στην Ελλάδα και αλλού. Πιστεύω πως ε, κάποια νέα προγράμματα για την καινοτομία αξίζει τον κόπο να τα εξεταστούν. Ας πούμε, στήριξη ε, διαφόρων ενώσεων φοιτητικών ε, στα πανεπιστήμια της Ευρώπης. Μεταρρύθμιση των πανεπιστημίων είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το μετακινηθούν από τα παλαιά πρότυπα στα πρότυπα της καινοτομίας είναι πολύ δύσκολο, χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Έχει γίνει συζήτηση για ένα κέντρο καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Silicon Valley. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποστηρίξει αυτές τι πρωτοβολίε και θέλω να ευχαριστήσω και, και να συγχαρώ την Επιτροπή σας που υποστηρίζει τη δημιουργία αυτού του κέντρου και τέλος να σας πω ότι δουλεύουμε με μέληψη στοιχείων, δηλαδή δεν γνωρίζουμε ποιε είναι οι επιπτώσει τη Silicon Valley για τη δημιουργία θέσεων απασχόληση εδώ στην Ευρώπη. Εγώ από διάφορα που ακούω θεωρώ πως άμεσα συμβάλλει η Silicon Valley δόση για τη δημιουργία θέσεων απασχόληση, αλλά χρειάζονται μελέτες για να το επικυρώσουμε αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τεράστιο αριθμό πληροφοριών που λάβαμε. Ας εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία να υποβάλουμε ερωτήσει τώρα. Δεν πρέπει να κάνουμε όλες τις συζητήσεις που κάνουμε στην Επιτροπή μας ούτως ή άλλως. Τι έχουμε τώρα, 40-50 λεπτά στη διάθεσή μας και μπορούμε να εμβαθύνουμε στις προφορές που πήραμε. Καταρχήν θα ήθελα να δώσω το λόγο στη συνάδελφο Μέρκης που είναι η συγγήτριά μας να ξεκινήσει εκείνη. Και όποιο άλλο θέλει να υποβάλει ερωτήσει ή να μιλήσει θα ζητήσει το λόγο θα το καταγράψουμε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε όλους τους ομιλητές μια που ήταν τόσο ενδιαφέροντα τα όσα μας είπαν στη σημερινή μας συζήτηση. Ορισμένοι εξημών ε, προκάλεσαν ιδιαίτερα με αυτά που είπαν και αυτό ήταν ε, σωστό για να η συζήτηση και ξεκινώ από τον τελευταίο από τους ε, αγορητάς και εσείς εάν κατάλαβα πάρα πολύ καλά μας είπατε ότι τα πανεπιστήμια μας είναι απειρχιωμένα είναι παλιωμοδίτικα Επομένως ε, μας λέτε ότι ε, δίνουμε περισσότερο τη σημασία στην ε, βασική έρευνα ενώ θα χρειαζόταν πιο εφαρμοσμένη πιο κοντά στην αγορά. Όμως αυτό οφείλεται και στο ότι τα περισσότερα πανεπιστήμια στην Ευρώπη δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε επιχειρήσεις venture capital, επιχειρηματικού κεφαλαίου και ε, ε, χρηματοδοτούνται και στηρίζονται και από τον κρατικό κορβάνα. Άρα, εσείς κύριε Σουμπλέ, για παράδειγμα, τι λέτε. Νομίζετε ότι έτσι θα μπορούσαμε να έχουμε την έρευνα πιο κοντά στην αγορά, εάν καταφέρουμε μια πανεπιστημιακή μεταρρύθμιση και έτσι να έχουμε μια συμμετοχή και του δυτικού κεφαλαίου στα πανεπιστήμια ο όμως πρόσβαση να έχει και η έρευνα στο ιδιωτικό κεφάλαιο. Άρα εκεί υπάρχει κάποιο κίνδυνο θεωρείται. Επίση κάτι άλλο. Μα είπατε ότι η Silicon Valley φτιάχνει θέσει εργασία, δημιουργεί θέσει εργασία. Τότε γιατί να μην κάνουμε και μια Silicon Valley και στην Ευρώπη. Και θα αποδώσει μόνο αν η προσέγγιση είναι παγκοσμιοποιημένη ούτω ή από όσο μας είπατε, μάλλον προσανατολίζεστε προς πρότυπα ασιατικά και όχι ευρωπαϊκά. Γιατί, μήπως θεωρείτε ότι τα ε, κατάλληλα απαραίτητα υλικά βρίσκονται εκεί και μόνος όλα αυτά τα οποία σπανίζουν τα, μπορούμε να τα βρούμε εκεί πέρα. Δηλαδή έχουμε τη δημιουργικότητα, αλλά δεν έχουμε το, την πρώτη ύλη. Και τα υλικά που γενικά. Επίσης μας είπατε ότι Εκεί είπατε ότι προχωράει περισσότερο καινοτομία παρά στην Ευρώπη. Γιατί γίνεται αυτό, κύριε Σουμπλά, μα είπατε ότι χρειαζόμαστε πιο ξεκάθαρα κριτήρια για το τι πάνε να πει καινοτομία στον τραπεζικό τομέα. Και όλοι είπατε ότι θέλετε ευελιξία, ε, ανοιχτό μυαλό, ελευθερία. Και αυτά τα κριτήρια δεν αντιβαίνουν σε αυτό το οποίο θέλουμε, δηλαδή στην ευελιξία το να έχουμε ακριβώ ξεκάθαρα σαφή κριτήρια. Το είπατε ότι είμαστε κάπως φορμαλιστές τυπολάτρες στην ε, Ευρώπη. Πιο πολύ ο τύπος μας ενδιαφέρει παρά το περιεχόμενο, άρα πώς μπορούμε να έχουμε περισσότερη πυρογνωμοσύνη που να βοηθούν τα προγράμματά μας. έχουμε καλύτερη συνεργασία με την ε, βιομηχανία. Και τελευταία ερώτηση. Στον κύριο Βασάρ. Εάν επικεντρωθούμε στην αποτελεσματική χρήση των πόρων τι θα κάνουμε και αν έχουμε πάρα πολλές από αυτές τις κοιλάδες που περιγράψατε ποιος θα αποφασίζει ποιες από τις κοιλάδες θα επιζήσουν προσέγγιση πρέπει να γίνει από πάνω προς τα κάτω Σας ευχαριστώ πολύ Επόμενη ερώτηση ο συνάδελφος Κύριε και αν ε, συμφωνείτε θα μαζέψουμε μερικέ ερωτήσει και θα σα απαντήσετε όλε μαζί. Εγώ ήθελα μόνο να κάνω μια παρατήρηση. Μετά από την παρουσίαση, ιδιαίτερα σε σχέση με τα όσα είπε ο κύριος από τη Φιλανδία. Τι, αυτό που σκέφτεται κανείς εδώ είναι Ποιος είναι ο λόγος για την έλλειψη, το χαμηλό επίπεδο της καινοτομίας. Εγώ πιστεύω πως η αγορά για την καινοτομία είναι μονοπωλιακή και αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Το μονοπόλιο θα πρέπει να καταργηθεί. Μεγάλες επιχειρήσεις κάποιες φορές μπλοκάρουν την αγορά παίρνουν ευρεσιτεχνίε που μπλοκάρουν άλλε πηγέ ε, ευρεσιτεχνία, καινοτομία και από την άλλη πλευρά οι μικρομεσαίε και οι ερευνητέ από τα πανεπιστήμια χρειάζεται να περιμένουν τρία-τέσσερα χρόνια μέχρι ότου εγκριθεί η ευρεσιτεχνία του. Και αυτό είναι το σημείο εκκίνηση. Εάν υπήρχε άλλο τρόπο, ε, σκέφτομαι α πούμε ένα ευρωπαϊκό γραφείο ευρεσιτεχνία, μάλλον μια ηλεκτρονική δυνατότητα χορήγηση ε, διπλώματος ευρεσιτεχνία δωρεάν ε, που θα υπήρχε και που θα μπορούσε έτσι να εγγυηθεί τα δικαιώματα των εφευρετών. Νομίζω πως τότε το κίνημα της καινοτομία θα αυξανόταν και θα ε, ενισχυόταν. Υπάρχει αυτό το βιβλίο ο αλγόριθμος της καινοτομία από έναν Ρώσο συγγραφέα που αποδεικνύει με βάση αλγορίθμους ότι οτιδήποτε μπορεί να εφευρεθεί. Αυτό το δυναμικό εφεύρεσης ε, στην, στην κοινωνία είναι πολύ ψηλό, αλλά δεν έχουμε, το έχουμε αντλήσει αρκετά. Γι' αυτό μου άρεσε τα όσα είπε ο ειδικό από τη Φιλανδία, γιατί μου είναι ιδιαίτερα προσφυλή και βλέπω πώς σκεφτόμαστε με τον ίδιο τρόπο. Ο συνάδελφος Οντί. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τις υψηλού επίπεδου εισηγήσεις σας. Εγώ είμαι εισηγητής για την αξιολόγηση και την αναθεώρηση του 7ου προγράμματος πλαισίου έρευνας και ανάπτυξης και επειδή το, οι προθεσμίες είναι πολύ σύντομες για τη διοργάνωση μιας ακρόασης θα εκμεταλλευτώ αυτήν την ακρόαση για να θέσω δύο-τρεις ερωτήσεις και να θυμίσω σύντομα το πλαίσιο η Κομισιόν είχε την υποχρέωση να κάνει την ανακοίνωσή της το 2010. Είναι τέσσερις ε, μήνες πίσω και δημοσιεύθηκε χτες. Σίγουρα δεν θα το έχετε διαβάσει κιόλας, αλλά σήμερα υπάρχουν δύο, τρία νέα στοιχεία. Το πρώτο είναι ο νέοι ναι, πολιτικοί θεσμοί που ορίστηκαν πέρυσι, ε, το 2009, νέα κομισιόν, νέο Ευρωκοινοβούλιο. Δεύτερο νέο στοιχείο είναι ότι έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε αποτύχει όσον αφορά τη στρατηγική της Λισαβόνας και γνωρίζουμε γιατί τα κράτη-μέλη δεν συντονίζονται με την Ένωση ούτε στην έρευνα, ούτε στις οικονομικές πτυχές, δεν υπάρχει στη σύμφωνη σταθερότητα κτλ. Και φτιάξαμε ένα νέο δικό χάρτη που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση 2020. Έπειτα, οικονομική κατάσταση. Το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο το διαπραγματευτήκαμε 2005-2006 και το ψηφίσαμε το τέλη 2006 για την περίοδο μέχρι το 2013. Δηλαδή, πολιτικώ αποφασίστηκε πριν την κρίση. Είμαστε στη μέση τη κρίση, πολύ ευαίσθητε ε, χρονιέ οι επόμενε και επομένων ε, το 11, το 12 και το 2013. Τα χρήματα που έχουν δαπανηθεί όμω και είναι μεγάλα ποσά Θυμίζω, πρόκειται για 51 δις ευρώ σε σύγκριση με το προηγούμενο πρόγραμμα πλαίσιο που ήταν 17 δις. Αυτά τα χρήματα συνήθως δαπανώνται στο τέλος των προγραμμάτων. Στα επόμενα χρόνια λοιπόν έχουμε ένα σώρο χρήματα για ευαίσθητα όμως χρόνια εξόδου από την κρίση. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν ε, μπορούν να αλλάξουν κάτι σε αυτό το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο γνωρίζοντας ότι στην αξιολόγηση της Κομισιόν γίνεται ένα είδος εξέτασης και copy-paste των όσων λένε οι εμπειρογνώμονες. Αλλά στην Κομισιόν δεν φαίνεται να υπάρχει αυτή η βούληση να κινηθεί Όλα όμω αλλάζουν το πάρα πολύ γρήγορα. Εμεί δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι άστα θα τα κάνουμε αυτά στο 8ο πρόγραμμα πλαίσιο που θα ξεκινήσει το 14, ενώ το 7ο ε, συνεχίζεται, τρέχει με σημαντικά ποσά. Κατά την άποψή σα, υπάρχουν πράγματα που πρέπει να μεταβληθούν στο 7, στο 7ο προ το συμφέρον τη Ευρωπαϊκή οικονομίας. Μπουτιέρες Κορτίνες. Ευχαριστούμε πολύ πάρα πολύ μεγάλη προσοχή σας άκουσα και θα ήθελα ε, να, το, να σας ξαναακούσω όπως κάνουμε τα έργα να σας ακούσω ξανά και ξανά συνέχεια Ολονύχτη. Λοιπόν, υπάρχει κάτι το οποίο εδώ πέρα με εντυπωσίασε, γιατί μιλάμε εδώ πέρα για την καινοτομία, όμω εδώ πέρα έχουμε και κάτι άλλο το οποίο είναι βαθύτερο, γιατί εδώ πέρα Υπάρχουν ε, πάρα πολλέ φιλοσοφίε που θα πρέπει να τι αναθεωρήσει κανεί, ούτω ώστε να μπορέσουμε να βρούμε έναν κοινό παρανομαστή. Ε, είναι, είναι κάτι το οποίο διαπνέει όλε αυτέ τι ομιλίε θα πρέπει να αλλάξει η συμπεριφορά, η νοοτροπία. Δηλαδή το πώ κανεί θεωρεί ότι πρέπει να δουλεύουν τα θεσμικά όργανα, η, η γραφειοκρατία, τα κράτη. Ε, και κάτι άλλο, νομίζω ότι υπάρχει το πρόβλημα του ότι η Ευρώπη έχει, είναι κάτι κάτι σαν σύνδρομο νομοθετικό, σύνδρομο κανονιστικό, το οποίο ξεκινά από μια σύλληψη σχεδόν θρησκευτική σε σχέση με το τι πάει να πει εξουσία. Δηλαδή έτσι κανείς νομοθετεί, νομοθετεί χωρίς καμία ευελιξία ε, για έναν κόσμο, για μια κοινωνία που αλλάζει, που είναι ευέλικτος. Και η Ευρώπη συμπεριφέρεται επομένως με τρόπο γραμμικό, ευθύγραμμο και το Πιο σημαντικό θεωρείται το η γνώμη του κράτους παρά η αγορά. Αλλά α, εγώ δουλεύω σε Επιτροπή Περιβάλλοντος και το REACH ας πούμε το πρόγραμμα ε, για τα χημικά ε, ε, προσπαθεί να ρυθμίσει τα πράγματα επί, επί τη βάση τη ύπαρξη αυτών των, χημικών ουσιών και όχι επί τη βάση του, του πώ παράγονται, τι Και επομένω ε, αυτό αποτελεί μια τροχοπέδη στην καινοτομία. Δεν βοηθάει. Να, επομένως, κυβερνούμε επί τη βάση, αρχών όμως η κοινωνία είναι περίπλοκη. Και αυτό γίνεται κάθε μέρα. Ας πούμε για τα, για τα λοιπάσματα. Τα ζενιοκτώνα. Όλα τα βάζουμε στο ίδιο καλάθι. Τι πάει να πει αυτό. Ότι υπάρχει μια νομοθεσία που ουσιαστικά αφορά τον Βορρά και όχι τον Νότο και οπότε έχονται τα αντίστοιχα, ε, τα αντίστοιχα έντομα και τι γίνεται, τώρα τις μέλισσες και σκοτώνονται τα, τα, τα, που πρέπει από αυτά τα ζένιοκτώνα. Προσπαθούμε να τα προβλέψουμε από πριν τρόπο ανελαστικό, να πούμε, για την αύξηση θερμοκρασίας. Θα πεθάνουν κάποια ζώα. Είδατε, θα, θα γίνουμε σαν την Αφρική από θερμοκρασία. Επομένω, χρειάζεται κάποιο είδου εξωτερική ε, συμβουλή ε, για να δούμε πώ θα μπορέσει να αλλάξει η κατάσταση. Δημιουργικότητα και καινοτομία εμποδίζονται με αυτόν τον τρόπο στην Ευρώπη. Άρα αυτό θα πρέπει να γίνει, να κάτσουμε για να ξαναδούμε τι γίνεται με τις αρχές μας, τι γίνεται εδώ στα θεσμικά όργανα. Επομένως νομίζω ότι αυτού του είδους η γραμμική νοοτροπία έχει σχέση με την περιπλοκότητα. Ε, θα πρέπει να προσθέσουμε τις μεθόδους μας, αλλά επίσης θα πρέπει να αναγνωρίσουμε την περιπλοκότητα. Επομένως, το γραφειοκρατικό κράτος δεν μπορεί να έχει την ίδια ταχύτητα όπως έχει η καινοτομία επιταχύνεται ο ρυθμός της καινοτομίας και αυτό το βλέπουμε κάθε μέρα. Α, στο facebook και άλλο. Άρα δεν είναι δυνατόν συνεχώς να βάζουμε όρια και όλα να υπάγονται στην έγκριση μιας γραφειοκρατίας. Άρα, να δούμε πώς λειτουργεί η εξουσία, πώς λειτουργούν τα θεσμικά όργανα, να ποια είναι η πρόκληση. Χρειάζεται τόλμη, χρειάζεται να κάνουμε κάτι το οποίο να σταματήσει να κατευθύνεται κατά τη κοινωνία. Συγγνώμη που είναι φορτισμένα ε, αυτά που σα λέω, αλλά νομίζω ότι τελικά η, ΦΙΕΝ, η κοινωνία είναι πολύ πιο έξυπνη, πολύ πιο ευφύ από ότι τα θεσμικά όργανα, από ότι εμεί. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Χέρτσοκ. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η μήνυα ακρόαση, Επομένω να πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια ε, τους συνεργάτες μας, τη γραμματεία, τον εισηγητή και όλου του συναδέλφου οι οποίοι προσήλθαν. Ε, τώρα έχω κάποιες ερωτήσεις και θα προσπαθήσω να είναι όσο είναι πιο στοχευμένες. Πρώτα-πρώτα, δύναμη της συνθήκης. Η, Ευρώπη, η καινοτομία κατέστη κοινοτική αρμοδιότητα. Όμως θα πρέπει να δούμε τι γίνεται σε επίπεδο κρατών, μελών και τι γίνεται σε κοινοτικό. τα κράτη-μέλη. Έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα, θα ήθελα να αποδιώξουν το συμπνικές αρμοδιότητες. Για ό,τι τουλάχιστον μπορεί να τα κάνει καλύτερα η Ευρώπη. Αν μπορείτε να μου απαντήσετε στο λίγο χρόνο που έχετε. Ε, ασχολούμαι πάρα πολύ με τις ΜΜΕ, έχω και μια σχετική έκθεση. Με λένε κυρία καινοτομία είναι το προσωνύμιο μου. Να δούμε όμω τι γίνεται με τι ευκαιρίε αυτέ. Τι ευκαιρίε υπάρχουν στα πλαίσια τη καινοτομία. Τι λέτε. Σε σχέση με το τι μπορούμε να πετύχουμε μέχρι τώρα, μέχρι πού έχουμε φτάσει. Πόσο μας απομένει ακόμα να καταφέρουμε σε σχέση με το δυνατότητά μας. τι μπορούμε να κάνουμε. Ανάλογα το τι μπορούμε να κάνουμε, λοιπόν, να διαλύσουμε και την κατεύθυνση στην οποία θα πάρουμε. Τώρα στη συνέχεια των όσων είπε ο Φιλανδός για την επέκταση. Ναι, η, η λιτότητα είναι καλή για τον προπολογισμό, αλλά, αλλά εάν έχουμε λιτότητα και στο μυαλό, στον προβληματισμό μας δεν πάμε μακριά. Άρα να τις συμβουλές. For SMEs. But just imagine how big problem we would have if the... Θα έπρεπε ΜΜΕ να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και να ξέρουν τι χρηματοδότηση μπορούν να βρουν. Αν ήταν έτσι τα πράγματα, δεν θα υπήρχαν μονοπόλια, γιατί και, το, και η πληροφόρηση έχει καταστεί μονοπόλιο. Επομένως, αυτό θα πρέπει να σπάσει. Να είναι γνωστό το χρηματοδοτικό πλαίσιο. Κύριε Οντή. Μακάρι να έβλεπα ε, όσο να βλέπω εσά και, και τον άντρα μου, γιατί είμαστε σε τρει επιτροπέ που συνεργαζόμαστε. Danke, Monsieur Keller. Kelly. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν, Δυστυχώ δεν άκουσα όλες τις παρουσιάσεις, γιατί ήμουν σε ένα σεμινάριο για την κοινωνία που είχε οργανώσει ε, η General Electric. Επίσης πριν από τα Χριστούγεννα Ήμουνα ε, τμήμα ελαβαμένο στην αντιπροσωπεία είπα ΕΕ και πήγαμε στην Αμερική και πήγαμε και στην ε, Silicon Valley. Είδαμε τι γίνεται εκεί. Όλες οι μεγάλες εταιρείε, eBay, Intel, ε, Intel, Google κλπ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τις ανάγκες που υπάρχουν για περισσότερη άλλη Δύο θέματα μας ενδιαφέρουν. Ο κύριος μας ε, προκάλεσε, γιατί εμείς δεν χρειαζόμαστε τίποτα άλλο παρά μια πρόκληση. Αναφερθήκε στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο και ότι δεν του επιτρέπεται ένα κριτήριο της ανάλυσης των ε, αιτήσεων να είναι η δυνατότητα εμπορίας. Αυτό είναι πεπαλαιωμένο νομίζω. Γιατί σε οποιαδήποτε προγράμματα χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίω για την έρευνα, θα υπάρχει έρευνα, ανάπτυξη και απόδοση. Η απόδοση είναι σημαντική. Και στις περισσότερε περιπτώσει θα πρέπει να είναι εμπορία. Αν υπάρχει λοιπόν ένα σφάλμα, εάν υπάρχει αποτυχία, εγώ συμφωνώ με την αμερικανική στάση. Καλύτερη αποτυχία παρά αδράνεια. Λοιπόν, πώς αντιδράει η Κομισιόν σε αυτά που τη είπατε εσεί και τι μπορούμε εμεί να κάνουμε για να φροντίσουμε ότι να αλλάξει αυτή η διάταξη. Επίσης μου φαίνεται πολύ προκλητικό και χρήσιμο ότι αναφέρονται σε πολλά από τα πανεπιστήμια δεν υπάρχουν στεγανά. Υπάρχουν ορισμένα πανεπιστήμια που λένε ότι είναι οι ηγέτες του κόσμου μέσα στους πύργους από ελεφανταστού που κάθεται. Ευτυχείς νομίζουν ότι κάνουν πολλά για τον κόσμο. Λοιπόν, θα πρέπει να ακούσουμε αυτές τις προκλήσεις και ελπίζουμε ότι θα υπάρχει μια αλλαγή. Και τι θα γίνει με τις αλλαγές αυτές στην Ευρώπη όσον αφορά τα πανεπιστήμια που δεν πρέπει να παρεμποδίζουν την καινοτομία, αλλά να τη διευκολύνουν. Είμαι σίγουρος ότι κάτι μπορεί να γίνει. Και χαίρομαι. Τα πανεπιστήμια ή να είναι προοδευτικά στο μέλλον ή να μην μας απασχολούν καθόλου. Να το αφήσουμε κατά μέρος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το Σνόφσκι. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα μιλήσω για να συμπληρώσω αυτό το οποίο άκουσα από του συναδέλφου, γιατί τα περισσότερα που άκουσα ε, με, με καλύπτουν. Θέλω να σα ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, διότι ε, σύμφωνα με είπα και ο Δόκτωρ Λί, ακούσαμε κάποια πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, κάποιες εναλλακτικές απόψεις σχέση με αυτό που ξέρουμε εδώ στην Ευρώπη και σε σχέση με αυτά το που γίνονται στη Silicon Valley και μας τα είπε κάποιο ο οποίο ξέρει τι γίνεται εκεί και αυτά έχουν σχέση και με το πρόγραμμα ε, εγώ κύριε Σαμπλέν έχω να σας ρωτήσω τα εξή. πώς θα καθοριστεί ποια εταιρεία είναι καινοτόμο και ποια όχι είναι πάρα πολύ δύσκολο διότι επί τη βάση τη εμπειρία μας εδώ στην Ευρώπη επί τη βάση των διαδικασιών που ισχύουν εδώ πάρα πολύ συχνά είναι δύσκολο να καθοριστεί αυτό και έχουμε ένα σωρό πράγματα, ε, προγράμματα εδώ και πολλές φορές ε, υπάρχει δυσπιστία. Οπότε και έχουμε όλη αυτή τη γραφειοκρατία, όλα αυτά τα έντια που πρέπει να Αυτό δεν θεωρείται ότι είναι ταφόπλακα για την γενοτομία και αυτό επίσης εμποδίζει το να καθοριστεί ποια εταιρεία είναι καινοτόμος και ποια όχι και πολλές φορές αυτό ε, δοκιμάζεται την ώρα που θέτει σε εμπορία η εταιρεία το προϊόν της, την υπηρεσία της. Κάτι άλλο κύριε Λί. Ε, είναι ένας συνάδελφος ο οποίος μας ανέφερε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά τα οποία θα πρικοδοτήσουν το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Εσείς ποιο θεωρείτε το πιο μεγάλο πρόβλημα γιατί εκεί θα κρυθούν πάρα πολλέ στρατηγικές, καινοτόμε και λοιπά. Όμως, για να είμαστε ειλικρινεί. Ε, το, εμπορικό πνεύμα είναι σχεδόν ύβρι στην ε, Ευρώπη. Όμως, αυτό είναι το σημαντικό τώρα, διότι για μας πολλές φορές είναι, είναι το, το εμπορικό πνεύμα, χαρακτηρισμός εμπορικός, είναι σαν κατηγορία, σαν κανείς να διαπράττει ένα δίκημα, σαν να κλέβει. Και έχουμε όλα αυτά τα ταμεία, τα περιφερειακά κλπ. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλές φορές ε, επικρίσεις ε, ότι ενώ έχει ε, κρατική ενίσχυση κάποιο τότε θα έπρεπε να έχει εμπορικό σκοπό. Μα τι γίνεται, εγώ ξέρω για κάποιο έργο το οποίο αξιολογήθηκε πρόσφατα. Πρόκειται για ένα συγκρότημα που θα βοηθήσει το Πανεπιστήμιο σε επίπεδο πληροφορικής και προσπάθησαν να αξιολογήσουν τις δυνατότητές του γιατί δύσκολο να αξιολογηθεί εάν εκεί θα γίνεται μόνο έρευνα. Και εφοβούνται, αν είναι δυνατόν, εφοβούνται ότι υπάρχει και εμπορικό στοιχείο. Οπότε αυτό είναι το θέμα ε, που, που, που ε, θα έπρεπε να σκεφτόμαστε ότι οποτεδήποτε και εμείς ίδιοι επενδύουμε χρήματα, φυσικά και θα έπρεπε, θέλουμε κάποια απόδοση. Άρα θέλουμε να έχει πιθανότητε επιτυχία κάτι μέσω αυτού του τρόπου. Ε, να πώ φρενάρει η καινοτομία. Τι λέτε. Τι λέτε. Μπα και πρέπει να αναθεωρήσουμε τα του 7ου ή του 8ου προγράμματο πλαισίου. Και θα πρέπει να εξορκίσουμε επιτέλους αυτό τον φόβο μας για την εμπορικότητα, τον εμπορικό σκοπό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, έχουμε λίγο ακόμα χρόνο, όχι πολύ, αλλά μπορούμε να ακούσουμε κάποιες απαντήσεις. Δεν θα μπορείτε όλοι να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Ο καθένας ίσως να συγκεντρώσει προσοχή σε κάποια ερώτηση για να έχουμε κατά δυνατόν πλήρες πληροφορίες ακόμα. Θα αρχίσουμε εδώ από τα αριστερά. Ο κύριος Σουμπλά. Ε, ε, Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δύο πτυχές που θα ήθελα να καλύψω. Η μεταφορά τεχνολογίας και σχετισμός μεταξύ πανεπιστημίου και έρευνας. Εδώ και 8-9 χρόνια πήραμε από τη Διεδική Διεύθυνση Έρευνας ε, κεφάλαια για μελέτη για να δούμε πώς θα υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποιήσει με αυτού του συσχετισμού. Δεν μπορεί τα δυνατόν να ε, αυτό μέσα στα πλαίσια του προγράμματος πλαισίου. Χρησιμοποιήσαμε άλλους πόρους, αλλά τότε είχαμε πάει στην Καλιφόρνια, στο Ισραήλ για να δούμε τι μοντέλα λειτουργούν και προσπαθήσαμε να καταλήξουμε σε κάποια λογική παρέμβαση. Αυτό όμως δεν είναι παντού δυνατό. Η μεταφορά τεχνολογίας προϋποθέτει δίπλα στο πανεπιστήμιο μια δομή χρηματοδοτική. Χρειάζεται δηλαδή μια ξεχωριστή νομική δομή όπου το πανεπιστήμιο θα είναι μέτοχος. και που θα ελέγχει το διαγωνισμό ανάμεσα στα πνευματικά δικαιώματα, τον έρευνα, το πανεπιστήμιο κλπ. Αυτό είναι μια ιδέα που είναι πολύ ανεπτυγμένη στη Σκανδιναβία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, λειτουργεί πολύ καλά, αλλά σε χώρε όπω και η Γαλλία έχουμε προβλήματα. Ε, και στην Ισπανία επίση αναζητείται μια λύση. Είναι πολύ πλοκό. Αν είχαμε περισσότερου πόρου, θα μπορούσαμε να τα αναπτύξουμε πιο συστηματικά. Χρειάζονται λοιπόν ειδικέ οικονομικέ ε, δομές δομέ γιατί δεν μπορεί άμεσα να επιδεθεί το κεφάλαιο στο Πανεπιστήμιο. Ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να αναφέρω η ανάγκη συνεργασίας και συνένωσης των προσπαθειών. Πολλές φορές αντιμετωπίζονται ε, κοινοτικές και εθνικές πολιτικές ε, που δημιουργούν κέντρα αριστείας, ε, κλάστερ, 80 ε, εδώ, 60 εκεί, 25 κάπου αλλού. δεν γίνεται αυτό. Χρειαζόμαστε 10-15 ε, τέτοιου τύπους κέντρα στην Ευρώπη. Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε από τόσα πολλά κέντρα προηγουμένης τεχνολογίας στην Ευρώπη. Ε, μια άλλη πτυχή, πτυχή. Εγώ είπα ότι θα πρέπει να είναι σαφής η ορισμή αλλά και ευέλικτη. Αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα και γι' αυτό το παλιό πρόγραμμα SIP τελικά στρέφεται προς τους πάντες. Γιατί δεν χρειάζεται να τίποτα. Πολύ πολύ πλοκό όμως το θέμα. Η κεντομία είναι ότι θα Μπορεί κάποια εταιρεία να ενταχθεί επειδή υιοθετεί κάποια και να τα διαδικασία. Επειδή εφευρίσκει κάποια καινοτομική διαδικασία. Τι ακριβώς. Θα πρέπει ο ορισμός να είναι σαφής. Γιατί εμείς είμαστε πρόσωποι της χοντρικής θα έλεγα. Δεν συνεργαζόμαστε άμεσα με τις επιχειρήσεις αλλά με τα τα μία με τις τράπεζες. Εμείς θέλουμε να υπάρχουν περισσότεροι πόροι, ούτως ώστε να μπορούν οι τράπεζες να κάνουν κάτι παραπάνω, τα ταμεία να κάνουν κάτι παραπάνω. Δεν έχουμε άμεση σχέση με τους πολίτες. Θα πρέπει δηλαδή οι τράπεζες να μην έχουν τον κίνδυνο να εναγκαστούν να επιστρέψουν ευρωπαϊκούς πόρους γιατί δεν είχε ακολουθεί το ακριβές σύστημα με την υποσημείωση που υπήρχε εκεί. Είναι πολύ άσχημο αυτό. Εγώ σημείωσα, συζήτησα με έναν υψηλό επίπεδο της Φινβερά, την Φιλανδία που είναι οι ηγέτες και είπε αυτά τα ευρωπαϊκά θέματα τόσο πολύπλοκα δεν θέλω καθόλου να ασχοληθώ. Και δεν χρησιμοποίησαν καθόλου το σύστημα αυτό. Είναι ακατανόητο. Πρέπει να υπάρχει σαφήνεια για τους ε, μεσάζοντες να υπάρχει απαραίτητη ασφάλεια να μπορούμε να συνεργαστούν με τα ευρωπαϊκά ταμεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και σα. Υπάρχουν διάφορε παρατηρήσει πολύ κέρυε που έγιναν. Ε, θα ήθελα εγώ να σχολιάσω το θέμα τη αξιολόγηση του προγράμματο πλαισίου. Φυσικά και τι εμπορικέ ε, πτυχέ και τι επιχειρησιακέ. Και επίσης πρέπει να μεριμνήσουμε για την επιλογή των αξιολογητών. Ε, πολύ ψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο. Ακτιμούμε τις γνώσεις τους, αλλά ποτέ δεν θα καταλάβουν όμως αν είναι πιθανή η εμπορία των αποτελεσμάτων. Άρα λοιπόν δική μου σύσταση είναι από τη μια πλευρά να αλλάξουν τα κριτήρια και να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε περισσότερο κόσμο που στοχεύει στη βιομηχανία κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης και από την άλλη πλευρά είναι ε, το θέμα του κατά πόσο υπάρχουν διαφορετικές δομές στην Ευρώπη. Την Ευρώπη, να σας πω όμως εγώ, δεν μπορούμε να την αλλάξουμε. Θα πρέπει να τη δεχτούμε όπως είναι. Να βρούμε όμως ιδέες για να ενισχύσουμε τη συνεργασία. Και αν δεν υπάρχει συνεργασία να επιτρέψουμε τον ανταγωνισμό. Και ας κερδίσει ο καλύτερο. Αυτό πρέπει να γίνει, να επιτραπεί και είναι κάτι που ούτω ή άλλω συμβαίνει. Φυσικά είναι απαραίτητη φυσικά και η προστασία ε, και η κάλυψη των κινδύνων γιατί διαφορετικά κανείς δεν θα τολμούσε να επενδύσει. Όμως θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος ποιότητος. Δεν μπορούμε δηλαδή να πηγαίνουμε από τη μια πλευρά στην άλλη. Να υπάρχει λιγότερη γραφειοκρατία, αλλά χρειάζεται σίγουρα έλεγχος ποιότητας. Κάτι άλλο που επίσης υπόθηκε είναι ότι από τη μια πλευρά ζητάμε και σαφή κριτήρια, από την άλλη πλευρά όμως χρειαζόμαστε, λέμε, περισσότερη ευελιξία. Και το θέμα ήταν κατά πόσο αυτό είναι αντίφαση. Όχι, δεν είναι αντίφαση. <clears throat> Και να σας δώσω ένα παράδειγμα από το ποδόσφαιρο. Έχουμε έναν απλό κανονισμό. Έχουμε 5-6 κανόνες, αλλά μεγάλη ευελιξία μέσα στο πλαίσιο του γηπέδου. Και αυτό χρειαζόμαστε και στην Ευρώπη. Ας πούμε, να ορίσουμε τις μεγάλες ε, προκλήσεις, τα θέματα στα οποία θέλουμε να εστιάσουμε την προσοχή, δηλαδή θα ήταν το γήπεδο, να έχουμε κάποιους βασικούς κανόνες και εσείς αναφέρατε ε, Μπέρτον πολλά κριτήρια που είπατε ότι πρέπει να υπάρχει λιγότερη κρατική ανάμεξη αλλά περισσότερο επιχειρηματικά κριτήρια, περισσότερη ευελιξία αυτό μετά να, να το γίνει. Να υπάρχει δηλαδή ένα συγκεκριμένο γήπεδο με συγκεκριμένους κανόνες. Και έπειτα αυτά που είπατε για τη Silicon Valley. Εγώ συμφωνώ για με τον Μπέρτον για όλα τα ωφέλη της Silicon Valley στην ΕΠΑ και έχουμε και εμείς αντίστοιχη προσπάθεια εδώ και ίσως και πιο ακόμα, πιο επιτυχή ακόμα αποτελέσματα στη Σανγκάη, στην Κίνα. Υπάρχει Silicon Valley στη Σανγκάη. Τώρα συζητάμε με τη ρωσική κυβέρνηση, με το Κόρκοβο, τη Silicon Valley της Ρωσίας, να δούμε πώς αυτό θα λειτουργήσει. Πολύ ενδιαφέρον το περιβάλλον. Εγώ λοιπόν αυτό που έχω να πω είναι ότι η Silicon Valley ως ιδέα είναι σπουδαία ιδέα. Μπορεί να γίνει και σε άλλα μέρη του κόσμου και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη πως διαφέρει το ένα μέρος από το άλλο. Υπάρχουν διαφορετικές κουλτούρες, νοοτροπίες. Μπορεί καν... Αυτό που ωφέλησε στη Silicon Valley είναι αυτή η νοοτροπία του να συγχωρεί κανείς την αποτυχία. Γιατί ακόμα και να αποτύχει κανείς στη Silicon Valley ε, θεωρείται ότι έχει εμπειρία. Ενώ στην Ευρώπη αν κάποιος αποτύχει θεωρείται ότι πάει, είναι χαμένος, αποτυχημένος. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή νοοτροπία όμως. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε πιο ανοιχτοί. Οι κανονισμοί εντάξει μπορεί να βοηθήσουν αλλά δεν το λύνουν το θέμα της νοοτροπίας. Σας ευχαριστώ. Just very briefly. Πολύ σύντομα. Εγώ εκπροσωπώ έψιλον Εταιρείε δηλαδή που βρίσκονται στην αγορά και θα ήθελα να πω ότι πραγματικά αυτοί που είναι στην αγορά, αυτό που χρειάζονται είναι την πρόσβαση στη χρηματοδότηση σήμερα, ίδιος ε, χρήματα για να ξεκινήσουν. Και ανησυχώ αν αυτό δεν επιληθεί, θα υπάρχει όσο πάει και λιγότερη κοινωνία στο μέλλον. Ιδίω αν πούμε ότι η ΜΜΕ είναι σημαντικό τμήμα τη αλυσίδα τη καινοτομία, γιατί πραγματικά αυτέ είναι που αναλαμβάνουν τον κίνδυνο. Χρειάζεται να υπάρχει όμω κάποιο κεφάλαιο γι' αυτό. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριο Σπάζαρη. Εκτός μικροφώνου. Υπήρξε μια ερώτηση από τον εισηγητή, ε, από την εισηγήτρια κυρία Μέρκης, για την πάρκια και κατά πόσο θα πρέπει να γίνει εκτίμηση από πάνω προς τα κάτω, από το κάτω προς τα πάνω. Εγώ αυτό που θα έλεγα είναι ότι πολλά από αυτές τις ε, κοιλάδες ε, όπως το Silicon Valley στην ουσία είναι σε χειμερία ανάρκη ε, και έχουν μόνο κάποιον που απαντά στα mail. Θα πρέπει να δοθούν κίνητρα, κάποιο είδος ανταγωνισμού για κάποια κριτήρια, κάποια κίνητρα. Αν, είσαι, αν πετύχεις, ας πούμε, θα ε, πάρεις το τάδε, βραβείο, διαφορετικά θα καταδικαστείς σε χειμερή ανάρκη. Οπότε θα ήταν και καλύτερο να κλείσουν. Αλλά φυσικά το να απαγορεύει κανεί τον κόσμο να προσπαθεί να αναλάβει πρωτοβουλία δεν είναι και το καλύτερο. Συνδυασμός δηλαδή τη φυσική επιλογή και των κινήτρων. Ευχαριστώ. So, last but not least, Mr. Lee. Τελευταίος ο κύριος Λί. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ ενθαρρυντικό είναι αυτό το οποίο άκουσα. Τη λέξη Facebook που είπαν οι ευρωβουλευτέ. Σα ευχαριστώ. Το χρησιμοποιώ. Το χρησιμοποιώ αρκετά. Πόσοι, πόσοι από σας μπήκα στο Facebook σήμερα. Α, μας σηκώνουν τα χέρια. Ωραία. Όλοι που δεν το έκαναν. Σας το συνιστώ. Αυτό του στα δίκτυα βοηθάνε επαγγελματικά. Το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ. Όλοι το χρησιμοποιούν το Facebook. Δεν είναι για τους teenager. Είναι για τους επιχειρηματίες, είναι για τις δουλειές. Ω, πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτό από το οποίο είπατε, είναι περίπλοκα τα θέματα. Ναι, ναι άκουσα ότι το εμπόριο είναι σχεδόν κάτι προκαλεί ανοχή. Υπάρχει και άλλη μια κακή λέξη από την άλλη μεριά του, του φάσματος. Ποια είναι η άλλη αυτή η λέξη που δημιουργείται. Έρευνα. Υπάρχει πάρα πολύ σκεπτικισμός, επιφυλάξεις, υποψίες στην βιομηχανία σε σχέση με το πώς γίνεται η έρευνα σε πολλά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Έχετε παγκοσμίου κλάσης πανεπιστήμια. Προσπαθούν να βελτιωθούν τα πανεπιστήμια γενικά στην Ευρώπη. Έχω, ε, έχω πολλά πανεπιστήμια και η έρευνα πώς γίνεται ενδιαφέρει πιο πολύ τους και όχι παραπέρα. Και είναι τα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, είναι τα θέματα της διάδοσης των αποτελεσμάτων της ερεύνης. Εάν δεν φτιάχτε σωστό πανεπιστημιακό σύστημα, τότε πάντα θα υπάρχει δυσλειτουργία όσον αφορά την έρευνα. Και αυτό δεν είναι για σας, αυτό είναι αρχή, παγκόσμια, ισχύει για όλα. Εκεί ακριβώς είναι το, η μεγαλύτερη τροχοπέδη για την καινοτομία. Είναι θέμα Ιαπωνίας, Ινδίας, Νοτιοαμερική. Θα πρέπει να αναθεωρήσετε τις θεμελιώδεις αρχές υπό των λειτουργούν τα πανεπιστήμια. Και αυτό είναι η ουσία του θέματος, της δυσκολίας της αλλαγής στην Ευρώπη. Γιατί οι αρχές σας ε, συγκροτήθηκαν, υιοθετήθηκαν τέλη του 19ου, αρχής 20ου αιώνα. Δηλαδή όπως είναι και και αλλού. Και αυτό γιατί θεωρήθηκε ότι βασικός των πανεπιστημίων είναι τον διδάσκει κανείς και ίσως παρεμπιπτόντω να κάνει και λίγο έρευνα. Στο Στάνφορντ και στο MIT, στο Μπέρκλεϊ και σε άλλα πανεπιστήμια, στο και όπω το Χάρβαρτ, κυρίω θέμα των πανεπιστήμιων είναι η έρευνα. Λέγονται ερευνητικά πανεπιστήμια. Και έτσι, έτσι κρίνονται όλοι. Καθηγητέ, φοιτητέ. Δημοσιεύσει που έχουν κάνει είναι βασικό. Οπότε η διδασκαλία των φοιτητών είναι σημαντική, αλλά δεν είναι αυτό που έχει την προτεραιότητα, το πρώτο. Όταν εσείς λοιπόν πρώτα-πρώτα προλαμβάνετε καθηγητές επί, επί τη βάση του πόσο καλά μπορούν να διδάξουν και όχι να κάνουν την έρευνα, τότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει μετά το πανεπιστήμιο και να αρχίσει να γίνεται ερευνητικό. Γιατί δεν έχει τους καθηγητές που, είναι, που έχουν καλές επιδόσεις σε αυτό στην έρευνα. Και αυτό με τη σειρά του κάτι που το έχετε κατοχυρώσει νομοθετικά. Δεν βλέπω να υπάρχει όμως προβληματική στην Ευρώπη όσον αφορά όλα αυτά. Για την αναθεώρηση αυτών όλων των προτύπων σας. Άρα, πρώτη θέση πρέπει να δώσετε στα πανεπιστήμια σας στον τομέα της έρευνας. Αλλιώς θα έχετε πρόβλημα. τη διοίκηση και τους καθηγητές που θεωρούν ότι πρώτο καθήκον είναι η διδασκαλία. Αυτή είναι η πρόκληση τώρα. Έχει αρχίσει βέβαια να αλλάζει η ισορροπία, μα και στην Κίνα, στη Λατινική Αμερική. Είναι βέβαια δεκαετίες πίσω, γιατί και εκεί ξεκίνησε με τη βάση δασκαλίας, ενώ οι Κινέζοι Τώρα είναι δεκαετίε μπροστά. Άρα θα ήθελα να Ευρώπη να ακούω περισσότερο όσον αφορά την, την αλλαγή τη ισορροπία. Γιατί αν αυτά όλα τα θεμελιώδη τα πετύχετε, τότε όλο το σύστημα θα βελτιωθεί. Πόση ώρα έχω. Άλλες παρατηρήσεις. Το Στάνφορντ. Όχι, δεν δέχεται επιχειρηματικό κεφάλαιο ιδιωτικό αλλά μη εμπορικό ίδρυμα είναι. Από την κυβέρνηση δίνονται υποτροφίες από ιδρύματα, από εταιρείε επίσης. Πληρώνουν διδακτρά. Αλλά υπάρχουν και λειτουργικές δαπάνες που καλύπτονται από τον προπολογό μας. Τρία δις δολάρια. Ένα δις είναι οι υποτροφίες που είπαμε ότι προέρχονται από εξωτερικά κεφάλαια. Όχι, άμεσα εμεί δεν συνεργαζόμαστε που είχαμε το κεφάλαιο. Οι δε εταιρείε που ιδρύουμε ή μάλλον εταιρείε με τι οποίε έχουμε σχέση η σχέση αυτή δεν είναι γραφειοκρατική. Αλλιώ δεν θα γινόντουσαν πολλά. Δεν θέλουμε να υπάρχει γραφειοκρατική διαδικασία και να περνάνε όλα πούμε, από τον πρίτανη. MIT, Harvard, σε όλα αυτά τα πανεπιστήμια εξετάζεται το τι εναλλακτικά μοντέλα υπάρχουν τόσο ώστε να πάμε προς την καινοτομία. Έρχονται πολλοί κόσμος να μας ε, επισκεφθεί, αλλά κανείς τελικά δεν ρωτάει το βασικό όσον αφορά την καινοτομία. Δηλαδή, τώρα το πτωχευτικό δίκαιο εδώ είναι το πρόβλημα. Να τον κανένα να τιμωρηθεί για πάντα, μπορεί να χάσει το σπίτι του, να τα χάσει όλα αν δεν πάει καλά η επιχείρηση. Και αυτό το οποίο κάνει η Ιρλανδοί σχετικά με αυτό θα πρέπει να γίνει κι αλλού στην Ευρώπη. Να κάνετε αλλαγέ. έτσι από την ε, αρχή της διαδρομής. Δηλαδή, αν κάποιος πήγαινε στην Μπακράτα δεν είναι δυνατόν να τιμωρείται όλη τη ζωή. Ακόμα και για τη μορφή της εταιρεία μιλώ. Όχι μόνο για ΜΜΕ, όπως κλασικά τις λέτε εσείς. Τώρα, οι στόχοι της ολοκλήρωσης Ευρωπαϊκής. Μήπως θα πρέπει να προσέξετε περισσότερο την εμπορική επιτυχία των ε, προγραμμάτων πλαισίων που έχετε, 7ο και το 8ο και να έχουμε... Βέβαια δεν είναι δυνατόν να έχει κανείς δημιουργία θέσεων εργασίας παντού το ίδιο γιατί ακριβώς το επιχειρηματικό κεφάλαιο είναι αλλιώς ε, η εμπειρογνωμοσύνη είναι αλλιώς κατανεμημένη, το κεφάλαιο αλλιώς και αυτό φέρνει εντάσεις βέβαια. Όταν ε, τα αποτελέσματα και η εμπορική επιτυχία των προγραμμάτων είναι άνηση, διαφορετική στη μία χώρα από την άλλη. Για κοιτάξτε, έχει προβλήματα δεν έχω τι απαντήσει, αλλά για κοιτάξτε. Α, Σανγκάη. Η Σανγκάη είναι ένα θύλακα πάρα πολύ σημαντικό, όλο ένα και πιο σημαντικό. Ναι, η Σανγκάη ανταγωνίζεται ή θα, πάρα πολύ γρήγορα θα ανταγωνίζεται τη Silicon Valley. Και η Ευρώπη είναι πολύ μακριά από αυτό το επίπεδο. Πάρα πολύ δύσκολο έτσι κι βέβαια να α, ξαναφτιάξει κανεί μία Silicon Valley. Ελάτε στο Στάνφορντ, επισκεφτείτε μας. Τι άλλο έχουμε. Άλλη μια βασική ερώτηση ε, θέμα το οποίο το ανέφερε η κυρία Γκουτιέρες Γκόμες, Κορτίνες. Τι θα κάνουμε με, την, με τον κόσμο που αλλάζει, οι αποφάσεις, οι εξελίξεις, οι επιταχυνόμενες. Αν η διαδικασία της αποφάσεων είναι κέντρο κατευθυνόμενη, μέσα σε αυτόν τον κόσμο που αλλάζει τόσο γρήγορα, τότε το μοντέλο αυτό μάλλον δεν είναι και τόσο καλό όσον αφορά την οικονομία και την ανάπτυξη. δεν είναι βιώσιμο ένα τέτοιο μοντέλο. Γι' αυτό και είναι τόσο αποκεντρωμένη η Silicon Valley. Από κάτω προς τα πάνω δουλεύουμε. Βέβαια, όσον αφορά την πολιτική για την καινοτομία, Έχετε κάποια να μου διδάξετε κι εσείς. Δεν είμαστε τόσο καλοί σε αυτό. Και πόσο αποδίδει τελικά η καινοτομία, τι, επιστροφή, τι απόδοση έχει το κεφάλαιο που κανείς έχει δώσει εκεί. Αυτό δεν είναι τόσο, δεν είναι τόσο βέβαιο. Δεν ξέρω. Από πλευρά θέσεων απασχόληση, κέρδου που προκύπτει, τι να σα πω. Αυτές είναι οι απόψεις μας. Έτσι πρέπει το πράγμα εμείς από τη Silicon Valley. Σας ευχαριστώ και πάλι. Πρόεδρος. Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους τους ε, εμπεριχνόμενες, την κυρία Μέρκης που τα προετοίμασε τόσο πολύ καλά. Ακούσαμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Αλλά πραγματικά μπορούσαμε κάπως να αισθανθούμε τι θα πει η καινοτομία. Σας ευχαριστώ γι' αυτό πάρα πολύ. Το τελευταίο λόγο έχει συνάδελφος Μέρκης. Σας ευχαριστώ ε, Πρόεδρο, ευχαριστώ τους ομιλητές ε, που ήρθαν εδώ, ευχαριστώ όλους τους παρόντες. Το κεντρικό θέμα ήταν ε, τι είναι η καινοτομία και ποιες είναι οι καινοτομικές ιδέες που επιτυχώς περνάνε στην αγορά. Ό,τι και αν είναι, θέλουμε πιο γρήγορα, πιο στοχευμένα, θέλουμε να κινηθούμε προς τις λύσεις και το θέλουμε στην Ευρώπη αυτό να γίνει. Χρειαζόμαστε λοιπόν καλύτερη αστίαση, καλύτερη χρηματοδότηση, περισσότερη σταθερότητα και απλούστευση. Και κυρίως χρειαζόμαστε φιλοδοξία. Χρειαζόμαστε αυτά τα σχέδια, τα μίνι Μανχάταν στην Ευρώπη και τον άνθρωπο που έφτασε στο, στη Σελήνη επίσης στην Ευρώπη. Και θα πρέπει να αλλάξουμε το ώστε να ενθαρρύνουμε την ε, δημιουργικότητα και γι' αυτό χρειαζόμαστε τόλμη. Χρειαζόμαστε τόλμη για να αφήσουμε το παρελθόν, για να πάρουμε αποφάσεις, για να εστιαστούμε, για να ορίσουμε αυτές τις μεγάλες προκλήσεις και το πώς θα φτάσουμε εκεί, με μια ελευθερία. Περισσότερες αυτές οι ιδέες ξεκίνησαν στο, μέσα στο σχέδιο έκθεση για την Ευρώπη της Καινοτομίας. Σας ευχαριστώ όλους που συμβάλλατε πριν από την ακρόαση και σας καλώ όλους να συνεργαστείτε και να περιοριστούμε στο διακανονισμό ο, της, ε, όχι της δημιουργικότητας αλλά της καινοτομίας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πέρα συνεδρίαση θα ξαναδοθούμε τέλη Φεβρουαρίου.